Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Parliaments, national governments. Να σας καλωσορίσω όλους. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους θερμά σε αυτή την ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, θα έλεγα στην Ευρώπη, αξιοσημείωτη γιατί, γιατί χρειαστήκαμε δύο χρόνια για να την προετοιμάσουμε. Την πρώτη φορά κανείς δεν είχε δηλώσει ενδιαφέρον από πλευρά ε, Εθνικών Κοινοβουλίων και των μόνιμων αντιπροσωπιών. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι τώρα πια ε, ευτυχώς τα καταφέραμε και χαιρόμαστε που ήρθατε. Έχουμε λοιπόν εκπροσώπους από 11 Εθνικά Κοινοβούλια και επιμελητήρια και έχουμε και τέσσερις προ ε, Προέδρους Επιτροπών εκπροσωπούνται η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Λετωνία, Κροατία, η Σλοβακία, η Γερμανία, Βέλγιο. Όλους εσάς λοιπόν σας καλωσορίζω θερμά. Ο συνάδελφος από την Εστονία λόγω της κυβερνητικής κρίσης ε, δυστυχώς δεν ήρθε. Το ίδιο ισχύει και για τον Πολωνό, ο οποίος δήλωσε ασθένεια. Αν δεν είχε συμβεί αυτό, θα είχαμε σήμερα περισσότερα, ε, περισσότερους εκπροσώπους και χειροσώματα που έχουμε τους μόνους εκπροσώπους μεταξύ αυτών την Κύπρο και άλλους Όλους εσάς λοιπόν σας καλωσορίζουμε. Για μας η ανταλλαγή απόψεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί η Επιτροπή Ελέγχου Προβλησμών ασχολείται με 80% το, του προβλησμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλαμβάνεται της κοινή διαχείρισης του περίφημου short management όπως λέγεται. Θέλουμε όμως να ακούσουμε και τη δική σας την άποψη και από την άλλη και εμείς επιθυμούμε να μεταφέρουμε το δικό μας το μήνυμα στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις. Και πάλι ευχαριστώ σας καλωσορίζω ή καλωσορίζω εκ μέρου του ελεγκτικού συνεδρίου τον κύριο Λαζάρου, ο οποίο είναι αρμόδιος για την περίφημη DAS, ε, τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος σε όλους τους τομεί του προπολογισμού. Αργότερα ο κ. Λαζάρου θα μας κάνει ε, τις ε, σχετικές του παρατηρήσεις. Και επίσης ε, ευχαριστώ και τον κύριο Τσέλερ, που ήταν αρμόδιο ε, για την απαλλαγή τη Κομισιόν του 2015. Ο κύριο Τσέλερ προέρχεται από το Βερολίνο. Θέλω να πω ότι για μα το ερώτημα το πώ ακριβώ χρησιμοποιούνται τα κονδύλια είναι ένα θέμα κλειδί. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε απλά να το ξεπετάξουμε, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, ε, όπω ε, θα μπορούσαν ίσω να πιστέψουν μερικοί. Δεν μπορούμε την χρήση των κονδυλίων να την πούμε ω κάτι το πεπατημένο που δεν μα ενδιαφέρει. Όχι, εμείς με τη χρήση των κονδυλίων επιτιμούμε να μαθαίνουμε συνεχώς για να γνωρίζουμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε ενδεχομένω του χρόνου. Καλωσορίζω λοιπόν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τον μόνιμο εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αγκρά, τον κύριο Μέγκελε, από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακά τον κύριο Μάρτιν και από τη Γενική Διεύθυνση Προεπολισμού τον κύριο Κραφ. Χαιρόμαστε που ήρθατε όλοι εσείς και ως εκ τούτου ε, θα κλείσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή στη συζήτησή μα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στου συζητητέ ε, για τον προπολογισμό του 2015. Επιτρέψτε μου επίση να επισημάνω ότι υπάρχουν και αυτά τα γαλάζια χαρτιά που κυκλοφορούν. Εκεί πρέπει να γράψετε το όνομά σα αν επιθυμείτε να λάβετε το λόγο. Και ε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να οργανώσουμε τη συζήτηση. Ο εισηγητή, ο κύριο Τσέλα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Λαζάρο, αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά, τα Περιφερειακά Κοινοβούλια και τι κυβερνήσει. Πρέπει να σας πω ότι και για μένα είναι πολύ σημαντικό το να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, γιατί πιστεύω ότι η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Περιφερειακών Κοινοβουλίων, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμεί στηρίζουμε ανεπιφύλακτα την περιφερειακή πολιτική. Αυτή λοιπόν η συνεργασία καθίσταται όλο και πιο σημαντική κατά τη διαμόρφωση των στόχων και κατά τη συμβολή μας για την επίτευξη των στόχων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε λιγάκι τα οικονομικά και μόνο τα οικονομικά. Δεν πρόκειται μόνο για την ε, απαλλαγή του 2015, γιατί πράγματι το 2015 είναι ένα ιδιαίτερο έτος, είναι δηλαδή το δεύτερο έτος στη νέα περίοδο στήριξης. Αυτό είναι το πρώτο. Από την άλλη όμως είναι και η πρώτη χρονιά όπου η νυν Επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες της. Αυτό το 2014 δεν είχε συμβεί. Η απαλλαγή για τον προϋπολογισμό κατ' ουσίαν σημαίνει και την έναρξη συζήτησης, ε, της ενδιάμεσης συζήτησης για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πρόκειται και επίσης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2017. Ξεκινάμε με τον ενδιάμεσο προϋπολογισμό όπως σας είπα, ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θα συζητήσουμε το τι θα γίνει με τα εργαλεία προαγωγής και στήριξης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να πω, ο ευρωπαϊκό προεκλογισμό σε μεγάλο βαθμό καταρτίζεται από τις συνεισφορέ των κρατών μελών, οι οποίες με τα οποία με τη σειρά τους καταβάλουν τις εισφορές εκείνες τις οποίες έχουν συγκεντρώσει από τους φορολογούμενους. Βεβαίως, η όλη αυτή η εφαρμογή είναι θέμα της εκτελεστικής εξουσίας, είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό όμως, κατά κανόνα, δεν εντάσσεται στους τοπικούς ή περιφερειακούς προϋπονολογισμούς. Παρόλα αυτά, εγώ θεωρώ, για να αναφέρω και να παραθέσω αυτά που είπε και ένας γνωστός Γερμανός Επίτροπος, είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα το 80% του ευρωπαϊκού προπλησμού όταν έχει εγκριθεί και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα δίλια αυτών επανέρχονται στα κράτη-μέλη και χρησιμοποιούνται για τη γεωργική πολιτική, για την ερευνητική πολιτική, για τα ερευνητικά προγράμματα, κυρίως όμως για την πολιτική συνοχή και για τα διαρθρωτικά ταμεία. Το γεγονός ότι τα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, αυτό είναι το ένα, πρέπει δηλαδή να εφαρμόζονται οι κανόνες που μόνοι μας έχουμε καθορίσει. Εξίσου όμως σημαντικό, αν θέλετε ακόμα και πιο σημαντικό, είναι η επίτευξη των στόχων οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί από κοινού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι να συμβαδίζουν με τα κονδύλια. Επ' αυτού λοιπόν έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Ακούμε όλο και περισσότερο ότι η επίτευξη των στόχων δυσχεραίνεται λόγω μιας συνεχώς διωγγούμενης γραφειοκρατίας. Υπάρχουν οι κανόνες ε, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη έχουν άλλους κανόνες και όπου οι περιφέρειες έχουν ισχυρή θέση, κατά κανόνα και οι περιφέρειες και αυτές ε, δημιουργούν τους δικούς τους τους κανόνες, πράγμα που σημαίνει τελικά ότι όσοι με διαδικασία εφαρμογής και εκτέλεσης, αυτοί έχουν πάρα πολλές δυσκολίες, απλά και μόνο λόγω του όγκου εργασίας ε, και όλων αυτών που οφείλουν να ε, επιτύχουν. Ως εκ τούτου, όταν καλούμετα να διεξάγουμε έλεγχο, αυτό βασικά είναι το καθήκον της Επιτροπής μας, εμείς εξαρτώμεθα από τα στοιχεία τα οποία μας δίδουν τα κράτη-μέλη. Στοιχεία, αξιολογήσεις, διαπιστώσεις και νομίζω ότι επ' αυτού και οι δυνατότητες του ελεγκτικού συνεδρίου είναι περιορισμένες. Άρα δηλαδή είμαστε αναγκασμένοι πλέον να συνεργαζόμαστε περισσότερο από ό,τι κατά το παρελθόν. Διότι νομίζω ότι έχουμε όλοι ένα κοινό στόχο, ένα κοινό διακύβευμα, το οποίο πρέπει και να εκφράζεται μέσα από τη συνεργασία μας. Εσείς που ασχολείστε με τα θέματα αυτά στα περιφερειακά κοινοβούλια αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια νομίζω ότι είναι χρήσιμο να συνεργάζεστε μαζί μας. Χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Θα έχουμε τρία πάνελ. Θα ακούσουμε διάφορες ε, διαπιστώσεις, ε, συμπεράσματα για το που έχετε καταλήξει εσείς και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την αξιολόγηση του προϋπολογισμού του 2015 αλλά και γενικότερα για το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με ευρωπαϊκές στρατηγικές ε, προγράμματα και με την εφαρμογή των κονδυλίων που θα σας διαθέσει ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στον πρώτο μιλτή, στον ε, κύριο Λαζάρου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παρακαλώ κύριε Λαζάρου, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζέλερ, για την απολογή του για την απαλλαγή του 2015 ξέρω ότι ήσασταν εισηγητή. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, όπω επίση και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν να ξεκινήσω ευχαριστώντα την ε, Προεδρία, όπω επίση ε, και ε, ε, την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών που μας κάλεσε να παρουσιάσουμε το θέμα αυτό. Για μένα πάντα αποτελεί μια ιδιαίτερη τιμή να μπορώ να παρίσταμαι σε αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμών και κυρίως παρουσία των τόσο αξιότιμων συμμετεχόντων και ομιλητών από τα εθνικά κοινοβούλια και από άλλους εθνικούς οργανισμούς. Είναι η πρώτη συνάντηση από τρεις που θα κάνουμε και θα λάβω το λόγο σε τρεις συνεδρίες. Θα ξεκινήσω λοιπόν κάνοντας μια πολύ σύντομη εισαγωγή στο τι είναι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε επίπεδο ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εμείς για τα θέματα προπολογισμού δεν λαμβάνουμε δικαστικές επαφάσεις, απλώς βοηθάμε στο να λειτουργεί καλύτερα μέσω των δικών μας εκθέσεων σχετικά με το θέμα αυτά και επικυρούμε, επικουρούμε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την, στην άσκηση του ελέγχου για την εφαρμογή του προϋπολογισμού. Μία από τις εκθέσεις είναι η ετήσια έκθεση για τους λογαριασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρουσιάζουμε μία χρηματοδότηση για την αξιοπιστία των λογαριασμών, όπως επίσης για την νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών. Εγώ είμαι επικεφαλής του πέμπτου ε, του πέμπτου τμήματος που έχει να κάνει με τις προσφυγές για θέματα ε, ε, ελέγχου του προϋπολογισμού και είμαι υπεύθυνο και για την ετήσια έκθεση. Στην σημερινή συνεδρία προσπαθούμε να βρούμε ένα νέο τρόπο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοίκηση των κρατών μελών. Και στην παρουσίασή μου θα ανατρέξω στο παρελθόν και θα δούμε ποιοι είναι οι ήδη υφιστάμενοι στόχοι του ελεγκτικού συνεδρίου της Ευρώπης έτσι ώστε να δούμε τι έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο καθόλου το διάστημα αυτό, έτσι ώστε οι δαπάνες να είναι λιγότερο δύσκολες, ε, λιγότερο, ε, περισσότερο ε, αποτελεσματικές και πιο εύκολο να ελεγχθούν. Τώρα για το 2016 είχαμε πει γύρω στα 140 δις ευρώ, είναι ο τρίτος ο χρόνος από το επταετές πολιτες πρόγραμμα για την περίοδο 2014-2020, οι δαπάνε μοιράζονται σε διαφορετικούς χώρους που είναι το πολιτες πλαίσιο και τα ε, κεφάλαια που ανήκουν σε αυτό. Τα κράτη-μέλη εμπλέκονται σε ένα μεγάλο βαθμό ε, στα θέματα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Θα ξεκινήσω λέγοντας από το γεγονός πως συλλέγουν και μοιράζουν τα περισσότερα έσοδα που στηρίζουν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Το Ελληνικό Συνέδριο υποβάλλει μια σχετική έκθεση στην πλαίσια της ετήσιας έκθεσης και επίσης έχει και κάποιες εξειδικευμένες εκθέσεις για παράδειγμα για το ε, ΑΕΠ και το 2013 και φέτος μιλήσαμε για το πώς, τι συμβαίνει σε επίπεδο ενδοκινοτικής απάτης για τον ΦΠΑ και δώσαμε κάποιες συστάσεις για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και στα κράτη-μέλη. Στα κράτη-μέλη οι αρχές επιλέγουν project και έργα για επενδύσεις, για να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής, για καλύτερη κατάρτιση, για να πέσει η ανεργία, όπως επίσης και για να πετύχουν υψηλότερε επενδύσεις. Τι κάνουν λοιπόν, ε, εξετάζουν και ελέγχουν τις αιτήσει πληρωμής των γεωργών όπω όπως επίσης και όσων συμμετέχουν στα προγράμματα συνοχής. Δηλαδή ε, ελέγχουν ουσιαστικά το 80% της κοινοτικής δαπάνης. Παρόλο που τον τελικό λόγο τον έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το 317 της συνθήκης, το ίδιο άρθρο αναφέρει πως ο προϋπολογισμός θα εφαρμόζεται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Και αυτό θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα η εξοικονόμηση πόρων να προσφέρει value for money και οι δαπάνες αυτές να προσφέρουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Έχουμε λοιπόν κάποιους μακρόπνους στόχους που ε, πλησιάζουμε σιγά σιγά και για την ονομοδότηση που είχαμε για τον ένα μοναδικό έλεγχο ε, συζητήσαμε το πώ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τι επιδόσεις μας στου ελέγχους και θα τα συζητήσουμε και στην τρέχουσα συνεδρία και στι ακόλουθε. Τώρα, στα ψηλά γράμματα να σα πω πω για να τα συνοψίσω όλα αυτά θα έλεγα. Πρέπει να διαχειριζόμαστε, να ελέγχουμε και να τεκπηριώνουμε τι δαπάνε με έναν ανοιχτό και διάφανο τρόπο, έτσι ώστε οι κοινοτικοί κανόνε να είναι απλοί, να είναι βανάγνωστοι, οι κανόνε αυτέ να στοχεύουν τι αναμενόμενε επιπτώσει και να μην έχουμε ε, αχρίαστη γραφειοκρατία. Θα πρέπει οι δαπάνε να ελέγχονται από τους ελεγκτές οι οποίοι βασίζονται σε τυχαία δείγματα έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να θεωρεί αξιόπιστη την προσπάθεια που γίνεται στους αρχικούς, στα αρχικά επίπεδα ελέγχου. Η φιλοδοξία μας είναι να εφαρμόσουμε αυτή τη single audit approach, δηλαδή την τακτική του ενός ενιαίου ελέγχου, μόλις πετύχουμε αυτά τα οποία επιδιώκουμε και πληρωθούν οι ε, προϋποθέσεις. Τώρα για το πρασίνισμα στα, στην γεωργία και για τις ενιαίες ενισχύσεις πρέπει να σας πω πως το υπολοιπόμενο ποσοστό σφάλματος έχουμε πετύχει καλύτερα ε, επίπεδα γιατί έχουμε οριμάσει. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Η παρακολούθηση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας βοηθά γιατί εσείς έχετε και τον τελικό λόγο στην παρακολούθηση του προπολογισμού αυτού και πρέπει να σας πω πως ο ρόλος σας είναι ιδιαίτερα σημαντικός και κυρίως η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού είναι ένας από τους βασικούς παίκτες μια και προετοιμάζει την έκθεση για την απαλλαγή που ψηφίζεται από την Ολομέλη. Όπως σας είπα και προηγουμένως, ένα μεγάλο κομμάτι της δαπάνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 80% ελέγχεται από τις αρχές των κρατών μελών. Και πρέπει να σας πω πως ε, εσείς βοηθάτε πολύ με τον τρόπο αυτό στην διαδικασία απαλλαγής στο ΕΚΟΦΗΝ, γνωμοδοτεί ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απαλλαγή. Άρα λοιπόν και τα περιφερειακά και τα εθνικά κοινοβούλια έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν, μεγάλο ρόλο γιατί εσείς εποπτεύετε τις δικές σας κυβερνήσεις και τις αποφάσεις για παράδειγμα για τα συγχρηματοδοτούμενα ε, ε, έργα στην στην συνοχή όπως επίσης και για τις γεωργικές επιδοτήσεις. Οι συνάδελφοί μου και εγώ θα βοηθήσουμε και το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Κοινοβούλιο σε αυτή την ε, λειτουργία της εποπτείας. Η ετήσια έκθεση δίνει το βαθμό αξιοπιστίας, μια γνώμη λοιπόν αξιοπιστίας για τους λογαριασμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την κανονικότητα των δαπανών όπως επίσης και των εισόδων. Οι συζητήσεις που γίνονται στα εθνικά και τα περιφερειακά ε, κοινοβούλια που γίνονται για θέματα δαπανών ε, έχουν πετύχει στο να επισπεύσουμε την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων ε, συνοχής και μας δίνεται και μια πιο πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει με τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες, είτε για γεωργικά θέματα, είτε για θέματα συνοχής. Ευχαριστώ πολύ, Μέγκελε, από την Επιτροπή Άγκρη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τον κύριο Λαζάρου. Θα ήθελα να συνταχθώ μαζί σου, να του πω πως χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε όλα τα επίπεδα τα οποία εμπλέκονται στις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία να συζητήσουμε μεταξύ μας, να βρούμε πού βρίσκεται το πρόβλημα και ίσως κάποιες ενδεχόμενες λύσεις. Όπως είπε μόλις και ο κύριος Τσέλερ, βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα, συνεισφέρουμε όλοι στα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο και βεβαίως με τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε όλοι να τα λύσουμε, κάτι το οποίο θα πρέπει να πετύχουμε με επικοδομητικό τρόπο. Τώρα, επιστρέφοντας στο θέμα της παρουσίασης που έχω να κάνω, οι λέξεις ε, εμπιστοσύνη και έλεγχος χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην ίδια φράση και ξέρουμε πως είχαμε ε, το, τη γνωστή φράση η ε, εμπιστοσύνη είναι καλή ε, αλλά καλύτερο ο έλεγχο και στην Wikipedia εμπιστοσύνη σημαίνει το να εμπιστευόμαστε κάποιον άλλον, άρα λοιπόν να δεχόμαστε τον έλεγχο που έχει κάνει κάποιο άλλος». Τι σημαίνει αυτό ότι ανοίγουμε και ένα παράθυρο στην αποτυχία αν ο εταίρος μας σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου δεν κάνει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να λέμε πως ο έλεγχος αποτελεί τη βάση της εμπιστοσύνης. Τότε προκύπτει το εξή ερώτημα. Πόσο έλεγχο χρειάζεται κανείς για να αποκτήσει αυτή την εμπιστοσύνη και πόση εμπιστοσύνη θέλουμε να δημιουργήσουμε εμείς μέσω αυτών των ελέγχων. Εγώ θα τα δω όλα αυτά από την πλευρά της ΚΑΠ και από, την, από κοινού ε, ευθύνη που φέρουμε, μια και είμαι ο Γενικός Διευθυντής που ε, έχει τον έλεγχο ενός μεγάλου κομμάτιου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η, ο βαθμός αποτελεσματικότητας της διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο της ΚΑΠ και των ελέγχων προκύπτουν σε κάποιο βαθμό από τα ποσοστά σφάλματος τα οποία βρίσκει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει να σας πω πως για την ΚΑΠ το ποσοστό σφάλματος είμαστε στο 2% που είναι λίγο πάνω από την ουσιαστικότητα, δηλαδή έχουμε αξιοπιστία για πάνω από το 97% των δαπανών που γίνονται στην ΚΑΠ. Για τον πρώτο πυλώνα, για τις άμεσες επενδύσεις και τα μέτρα αγοράς, είμαστε στο 2,2% ποσοστό σφάλματος, το οποίο είναι σχεδόν σε επίπεδο ουσιαστικότητας, ενώ για το δεύτερο πυλώνα δυστυχώς είμαστε ακόμα στο 5,3%, το οποίο σημαίνει πως ακόμα χρειάζονται να γίνουν μεγάλες βελτιώσεις. Όμως, όταν εστιάζουμε στους συγκεκριμένους οργανισμούς πληρωμής, θα δούμε πως η εικόνα που αποκομίζουμε είναι αρκετά διαφοροποιημένη. Για να δούμε τι ήταν η αξιολόγηση στην ετήσια ε, δική μας έκθεση για τον δεύτερο πυλώνα που κάναμε στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Είχαμε επιφυλάξεις εδώ για 24 οργανισμούς πληρωμών γιατί ήταν πάνω από το 2% και δεν είχαμε αρκετά ελαφρυντικά στοιχεία για να το εξηγήσουμε. Όμως αυτό σημαίνει ότι οι 48 οργανισμοί πληρωμών ήταν είτε κάτω από την ουσιαστικότητα είτε τουλάχιστον δεν χρειαζόταν επιφύλαξη για τη δράση τους. Η DG Agri, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, κατέληξε σε αυτούς τους υπολογισμούς λόγω των δικών της διαδεδομένων, πολύ διαδεδομένων ελέγχων και χρησιμοποιώντας και άλλες πηγές ελέγχους όπως για παράδειγμα και το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και οι φορείς πιστοποίηση των κρατών μελών. Αυτό αποδεικνύει ότι η αξιοπιστία για να είναι πραγματική και αν αυτή γραμμίζεται με τα όσα λέει ο κανονισμός δεν μπορεί να προσφέρεται χωρίς να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα ελεγκτικής δραστηριότητας και για την αξιοπιστία των ελέγχων και των δεδομένων που στέλνουν οι οργανισμοί πληρωμών στην DG Agri, πρέπει να πούμε πως είναι αξιόπιστα τα στοιχεία αυτά, στο βαθμό που δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρούμε πως τα κράτη-μέλη θα μας έστελαν λανθασμένα ή χειραγωγημένα στοιχεία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως οι υποκείμενοι έλεγχοι, οι οποίοι γίνονται από τους οργανισμούς πληρωμών, σε πολλές περιπτώσεις δεν ανοιχνεύουν όλα τα σφάλματα ή τις παρατυπίες οι οποίες διαπιστώνονται επί Και για το λόγο αυτό η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας όταν υπολογίζει στην έκθεση τη δραστηριότητα στο ποσοστό σφάλματος προσαρμόζει τα δεδομένα ελέγχων που στέλνουν τα κράτη-μέλη προ τα πάνω, χρησιμοποιώντα όλες τις πληροφορίε που έχει για ελέγχου και Όσο πιο πολύ συχνά οι φορείς πιστοποίησης δίνουν στέρεες γνώμες για τη δουλειά του οργανισμού πληρωμών, τόσο, πολύ, τόσο πιο πολύ μπορεί η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας να χρησιμοποιήσει αυτές τις πιστοποιημένες γνώμες στη δική της, στους δικούς της υπολογισμούς, μια και εξυπηρετούμε τα ίδια συμφέροντα που εξυπηρετεί και το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο, που είναι να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν σε αυτό το ε, έναν και ενιαίο έλεγχο. Η έλεγχη και η πιεστική αυτή έλεγχη για τους δικαιούχους και για τους οργανισμούς πληρωμών πληρωμών πολλές φορές επικρίνονται και μας λένε πως είναι υπερβολικός ο αριθμός και δημιουργεί ε, διοικητικό βάρος. Και πρέπει να σας πω πως υπάρχει μια μειωμένη ανάληψη μέτρων ΚΑΠ ε, λόγω ακριβώ του διοικητικού βάρους αυτός. Κοιτώντας αυτές τις επικρίσεις πρέπει να δούμε πως στοχεύουν σε δύο τελείως διαφορετικά μεταξύ τους φαινόμενα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είναι περίπλοκη η πολιτική. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακούγεται συνέχεια για τα στοχευμένα κομμάτια της ΚΑΠ και πιο συγκεκριμένα για το δεύτερο πυλώνα. Και δεύτερον, ότι είναι πολύ βαρύ το φορτίο των ελέγχων και των κυρώσεων σε επίπεδο δικαιούχων και μας λένε πως είναι υπερβολική και πολύ εντατική η έλεγχη που γίνονται στο πώς κάνουν τις δαπάνες στους οργανισμούς πληρωμών. Να σας πω λοιπόν πως το δίλημα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με όλα αυτά είναι το εξή. Πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε το διοικητικό βάρος που προκύπτει από τους ελέγχους και παράλληλα να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε χαμηλά επίπεδα ασφάλματος και μια εφαρμογή της ΚΑΠ θα είναι αποτελεσματική από πλευράς κρατών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά, θα ήθελα να σας δείξω τι κάνουμε και να συζητήσουμε τους τέσσερις βασικούς λόγους για τους οποίους ενεργοποιούμε ελέγχους και ελεγκτική δραστηριότητα. Πρώτα απ' όλα, να σας πω πως αποτελεί ε, κοινή παραδοχή πως η περιπλοκότητα των ελέγχων έχει να κάνει με το πόσο περίπλοκα είναι τα μέτρα τα οποία ελέγχουμε. Δηλαδή, το να μειώσουμε τον έλεγχο και το βάρος των ελέγχων σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε το πόσο περίπλοκη είναι η ΚΑΠ. Δηλαδή, απαιτεί απλούστευση. Ο Επίτροπος κ. Χόγκαν έχει προσπαθήσει να πετύχει κάτι τέτοιο από την αρχή της θητείας τους, εφαρμόζοντας μία σειρά από αλλαγές πλούστευσης στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, έχει αναλάβει να εξυγχρονίσει και να πλουστεύσει την ΚΑΠ σε βασικές πράξεις στα πλαίσια του πολυνομοσχεδίου, που το Omnibus, δηλαδή το πακέτο αυτό, το οποίο θα κατατεθεί στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό δεν είναι φιλόδοξο, γιατί τι μας αποδεικνύει η εμπειρία, πως η νομοθετική διαδικασία και η πολιτική διαδικασία λήψη αποφάσεων ουσιαστικά πολύ σπάνια έχει θέσει την απλούστευση ως προτεραιότητα. Α δούμε λοιπόν ποιο θα ήταν το ευκταίο επίπεδο συμμόρφωσης που αυτή τη στιγμή έχουμε θέσει ως το 98%. Αν Αναμφίβολα το να πετύχουμε αυτό το επίπεδο συμμόρφωσης αποτελεί έναν βασικό λόγο για τον οποίο έχουμε οδηγηθεί σε σκληρούς ελέγχους επιτόπου, σε εξαντλητικούς ελέγχους από πλευράς κομισιών και σε μια στενή παρακολούθηση. Και αυτό ισχύει κυρίως για τον πυλώνα 2 που έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό σφάλματος. Με μια συμφωνία η οποία ε, ζητά καλύτερο κατόφλι ουσιαστικότητας ε, που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις φιλοδοξίες που έχει η πολιτική μας, λέμε πως ακόμα τα ποσοστά σφάλματος θα πρέπει να ε, εμφανίζονται ε, με έναν τρόπο που θα μπορούν να διορθώνονται από ε, την Κομισιόν. Και στην έκθεση του 2015 δείξαμε πως για το γεωργικό χώρο στην στιγμή του κλεισίματος ο κίνδυνος είναι πάνω από την ουσιαστικότητα, ε, κυρίως αν λάβουμε υπόψη και τους επόμενους οικονομικούς καταλογισμούς, δηλαδή τις μελλοντικές διορθώσεις. Επίσης, διορθωτικοί μηχανισμοί σε επίπεδο κράτους μέλους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιούμε όπως μπορούμε τη νέα τεχνολογία και τις λύσεις που μας δίνει η πληροφορική. Η ολοκληρωμένη ε, διαχείριση του ΟΣΔΕ ε, μέσω του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμοχίων, το LPIS, και την διαδεδομένη χρήση της τηλεπισκόπησης, το οποίο σημαίνει ότι πια δεν γίνονται κλασικοί επιτόπιοι έλεγχοι, όπως επίσης και η εισαγωγή ενός νέου γεωστατικού ε, συστήματος και γεωχωρικού συστήματος που χρησιμοποιούν οι γεωργοί, μας οδηγούν σε ένα νέο σχήμα που μπορούμε να κάνουμε τους ελέγχους επιτόπου από μακριά και παράλληλα τα ποσοστά σφάλματος να παραμένουν χαμηλά. Με τον ίδιο τρόπο θα έπρεπε σε όλου του χώρου της ΚΑΠ να μάθουμε από την εμπειρία που μας έχει διδάξει ο ΩΣΔΕ και να δούμε πού στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε δεδομένα που είναι ε, ανοιχτά και όπου μπορούμε να κάνουμε ένα pre-screening των αιτήσεων έτσι ώστε στην προεκτυπωμένη αίτηση να μπορούμε να διορθώσουμε κάποια σφάλματα πριν αυτά κατατεθούν. Επίσης, ο έλεγχος που ειναι ανοιχτα και οπου μπορουμε να κανουμε ενα pre screening των αιτησεων ετσι ωστε στην προεκτυπωμενη αιτηση να μπορουμε να διορθωσουμε καποια σφαλματα πριν αυτα κατατεθουν επισης ο ελεγχος που βασιζεται σε αναγνώριση κινδύνου ε, που έχει να κάνει με την αρχή κόστους-οφέλους πέραν των υποχρεωτικών χρήσεων της ανάλυσης κινδύνου στον σχεδιασμό των επιτοπίων ελέγχων, οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των ελέγχων ε, για τις άμεσες ενισχύσεις από το 5% στο 3% και ίσως και στο 1% αν τα συστήματα ελέγχου που εφαρμόζουν λειτουργούν σωστά. Αυτή τη στιγμή έξι οργανισμοί πληρωμών χρησιμοποιούν αυτή την εναλλακτική που προσφέραμε και για το μέλλον η εναλλακτική αυτή ενδεχομένως θα μεταφερθεί και σε άλλα καθεστώτα έτσι αρκεί, αρκεί οι φορεί πιστοποιητή στη γνωμοδότησή του για την νομικότητα και κανονικότητα των πληρωμών αποδεικνύουν πω τα εθνικά συστήματα είναι αξιόπιστα. Και από αυτή τη βάση η Γενική Διεύθυνση Γεωργία, DG Agri, θα μπορέσει να επαναπροσανατολίσει τι ελεγκτικέ δραστηριότητε και να στοχεύσει περισσότερο στου οργανισμού πληρωμών με τον υψηλότερο κίνδυνο για παράτυπη δαπάνη. Τι σημαίνει αυτό, το να πλησιάσουμε περισσότερο την αρχή αυτή του single audit, της, του ενιαίου και μοναδικού ελέγχου που θα κάνουν του ελέγχου μα πιο αποτελεσματικού, και πολύ πιο στοχευμένους. Θα ήθελα τέλος να μοιραστώ μαζί σας κάποια πολύ προσωρινά συμπεράσματα για το πώς θα απλωστεύσουμε το νομικό πλαίσιο για την αγροτική ανάπτυξη πέραν του 2020. Ευθυγραμμιζόμαστε λοιπόν με την λογική που λέει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να εστιάζεται στα αποτελέσματα αυτού, στο μέλλον θα πρέπει να ε, επιδιώκουμε να πετυχαίνουμε προ προσδιορισμένους στόχους και αποτελέσματα και όχι τόσο πολύ να θέλουμε ε, τη συμμόρφωση με τις μυριάδες κριτηρίων επιλεξιμότητας. Άρα λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να διοργανώνονται ε, στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας και θα πρέπει στα μελλοντικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης να ευθυγραμμίζονται με τους νέους στόχους και τις νέες προτεραιότητες. Με ένα τέτοιο πλαίσιο η συμμόρφωση σε επίπεδο δικαιούχου θα μπορούσε να ε, μειωθεί και να περιοριστεί στο να έχουμε χρηστή οικονομική διαχείριση και κατάλληλες διαδικασίες. Βεβαίως, θα πρέπει να έχουμε κανόνες περί συμμόρφωσης, κάποιους βασικούς κανόνες που θα εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι. Για παράδειγμα, για κάποια θέματα α, ε, της αγροτικής ανάπτυξης, όπως επίσης, για παράδειγμα τα γεωργοπεροβαντολογικά ή κάποιους άλλους περιορισμούς, του ε, ε, ε, τους οποίους θα πρέπει να σεβαστούμε πριν επιδοτηθεί κάποιος. Ο υποπτικός ρόλος λοιπόν ο δικός σας θα έπρεπε να εστιαστεί σε δύο χώρους. Πρώτα απ' όλα στο να πετυχαίνουμε αποτελέσματα και στον έλεγχο των ευρωπαϊκών κανόνων. Γιατί αν έχουμε κάποιους νομικούς, ε, νομικά επιβεβαιωμένους στόχους απόδοσης στους δικαιούχους, τότε τι θα κάνουμε. Ένα, θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι πάρα πολύ απλό, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να αξιολογείται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Και εμείς θα δούμε μόνο τους ελέγχους ε, που ε, θα αξιολογούν το κατά πόσο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τα προγράμματα με αποτελεσματικό τρόπο και κατά πόσο σέβονται το απλουστευμένο νομικό πλαίσιο σε συμμόρφωση με την ε, εξάντερη με τον προληπτικό έλεγχο δηλαδή. Άρα λοιπόν, για μετά το 2020 υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε για την ΚΑΠ και αν πετύχουμε θα μπορέσουμε να μειώσουμε το βάρος των ελέγχων για τους δικαιούχους και σε επίπεδο οργανισμών πληρωμής. Όμως, για ένα σύστημα που βασίζεται στις αποδόσεις, η απλούστευση που μπορεί να γίνει τελικά θα σχετίζεται με το επίπεδο αξιοπιστία που θα ζητάμε από τους εξωτερικούς ελεγκτές ε, που ελέγχουν το πώς διαχειριζόμαστε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και αυτό θα περιορίσει ε, το, τη δυνατότητα εμπιστοσύνης που θα έχουμε στα κράτη-μέλη έτσι ώστε αυτά να εξασφαλίζουν τη χρηστή διαχείριση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε σε λίγο με τη λίστα των ομιλητών, με τον Υπουργό Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Αξονίας, τον κύριο Σμιτ. Χαιρόμαστε που, που βρίσκεστε εδώ. Όσον αφορά το θέμα, καλή εμπιστοσύνη αλλά καλύτερο ο έλεγχο. Να δώσω κάποιου αριθμού. Στην αγροτική ανάπτυξη η Σαξονία έχει ένα ποσοστό σπάλματος 2,76%. Αυτό ανέφερε προς τις Βρυξέλλες όπου και διορθώθηκε στο 4,4%. Ωστόσο, αυτό όσον αφορά το θέμα της εμπιστοσύνης και του ελέγχου. Για μας την... το ζήτημα του πόσο αξιόπιστα είναι τα στοιχεία που δίνουν στις Βρυξέλλες στα κράτη-μέλη είναι αποφασιστική σημασία. Επειδή μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Αν μπορούμε να βασιζόμαστε στους αριθμούς αυτούς, θα ήταν μια διευκόλυνση για εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε η δυνατότητα να παρουσιάσω εδώ τις ιδέες μας για την προώθηση της αγροτικής παραγωγής μετά το 2020 και τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις είχαμε αυτή την προσέγγιση, η οποία διαφέρει από τη δική μας. Κάποια λίγα λόγια για το δικό μας ομόσπονδο κρατήδιο, το ελεύθερο κράτος της Αξονίας. Είμαστε ένα από τα νέα ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Όπως είπατε, εποφελούμαστε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία 25 χρόνια από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Χωρίς αυτή την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάπτυξη του ελεύθερου κράτους της Αξονία, την οποία βιώνουμε τα τελευταία 25 χρόνια, δεν θα ήταν δυνατή. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη για μας. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη για τι περιφέρειες των χωρών που προσχώρησαν αργότερα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό για μας να διαμορφώσουμε διαδικασίες οι οποίες σε τελική αναλύση θα μπορούν να εφαρμοστούν στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι μία από τις προσεγγίσεις μας. Αλλά αρχικά θέσαμε το ερώτημα. Εάν πριν από κάθε μεταρρύθμιση ή κατά διάρκεια κάθε μεταρρύθμισης μιλούμε για απλοποίηση, γιατί είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί. Πιστεύω ένας λόγος είναι πως εάν μιλούμε μόνο για λεπτομέρειες εντός του συστήματος, τότε θα επιτύχουμε μερικές απλουστεύσεις, αλλά κατά την επικοινωνία των επιμέρους των τομέων μπορούμε να περιπλέξουμε και τα πράγματα. Γι' αυτό και η προσέγγιση μας έγκυται σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και όχι σε τροποποίησεις δευτομεριών. Και φυσικά πάντα βιαζόμαστε πολύ να αρχίσουμε συζητήσεις περιεχομένου για τις κατευθύνσεις της χρηματοδότησης. Δηλαδή πώς, ποια ποσά από τον προϋπολογισμό θα πάνε στη γεωργία, στην προστασία του περιβάλλοντος και σε άλλους επιμέρους τομείς και εκεί έχουμε τις πιο αμφιλογόμενες συζητήσεις. Γι' αυτό και εμείς την πρότασή μας, διαχωρίσαμε την πρότασή μας για την εφαρμογή του περιεχομένου ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα πάει στην προστασία του περιβάλλοντος ή σε άλλους τομείς. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε αργότερα. Για να επιτύχουμε την αποδοχή και μια λύση. Το είπαν και οι προλαλήσαντες Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο που θα μπορεί να εφαρμοστεί για νομικές τροποποιήσεις και για χρήση κονδυλίων. Με λίγα λόγια χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο το οποίο σε τελική ανάλυση θα μπορεί να εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη και θα μπορεί να τηρηθεί από τα κράτη-μέλη. Για μας, αναμφίβολα, η απάτη πρέπει να καταπολεμείται με σαφείς κυρώσεις, δεν το συζητούμε αυτό αλλά θέλουμε ένα διαχωρισμό της θεώρησης διαδικαστικών σφαλμάτων και, εκπρο... και εκπροθέσεως απάτης. Γι' αυτό και είναι σημαντικό για εμάς να επιτύχουμε την αποδοχή της Ευρώπης σε αυτόν τον κόσμο που τόσες αναταραχές βιώνει σήμερα και να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη. Αυτό πιστεύω πως μας ενώνει όλους. Ε, οπτικοποιήσαμε το πλαίσιο των κανονισμών, των λαβύρινθων αυτών των κανόνων που πρέπει να τηρούμε. Αρχίσαμε το 1994 με έναν κανονισμό 80 σελίδων, ένα πρόγραμμα με 80 σελίδες, τρεις κανονισμοί από 30 σελίδες η καθεμία και ένα σχέδιο με χίλιες σελίδες και 24 κανονισμούς με ένα σύνολο σχεδόν αρκετών χιλιάδων σελίδων όγκου. Εδώ έχουμε το πρώτο πρόβλημα. Αν θέλουμε να τα τηρήσουμε όλα αυτά, αν σε κάθε έλεγχο έχουμε τέτοιους κανόνες, τότε τα σφάλματα στη διαδικασία είναι αναμενόμενα. Ακόμη και αν έχουμε μια πολύ εξειδικευμένη διοίκηση, στο τέλος δεν μπορούμε να τηρήσουμε όλες αυτές τις προδιαγραφές. Γι' αυτό και τα προβλήματα είναι αναμενόμενα για τις διοικήσεις των κρατών μελών και των περιφερειών τους. Γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο προλαλήσαντας μίλησε, έθιξε το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό να επιτυγχάνεται ο στόχος στο τέλος. Αποφασιστικό δεν είναι εάν η ταμπέλα που βρίσκεται πριν από το μέτρο χρηματοδότησης είναι 2 3 εκατοστά μεγαλύτερο ή μικρότερο. Επειδή αυτό το ε, σπάλμα μπορεί να διορθωθεί στο τέλος, αλλά δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με κυρώσεις. Το ελεγκτικό σύστημα θυχθήκε επίσης. Πλέον έχουμε ένα σύστημα ελέγχου από την οπτική γωνιά της Σαξονίας, στο οποίο συμμετέχουν 12 θεσμοί και πολλές φορές τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα ενιαίου ελέγχου και πρέπει να καταρτήσουμε σαφείς κανόνες για το ποιο είναι αρμόδιος για ποιον έλεγχο. Το άχθος που κρύβεται πίσω από αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το ελεγκτικό συμβούλιο της Βάδης Βιρτεμβέργης υπολόγισε για την τελευταία περίοδο όταν το άχθος δεν ήταν τόσο μεγάλο πως ξοδεύονταν 100 ευρώ για την για τον καταμερισμό 300 ευρώ χρηματοδότηση. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Υπήρξε και ένα ακραίο παράδειγμα στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν 9.000 ευρώ για να διαπιστωθεί ένα σφάλμα ύψους 23 ευρώ. Αυτός πιστεύω πως είναι ο λάθος δρόμος. Και εμείς στο ελεύθερο κράτος της Αξονίας μπορούμε να αναφέρουμε παραδείγματα, πολύ σύντομα ένα, λόγω ενός τυπικού σφάλματος για μια χρηματοδότηση για μια χρηματοδότηση 3.500 ευρώ προκάλεσε δαπάνες 860.000 ευρώ στο ελεύθερο κράτος της Αξονίας. Αυτό σημαίνει πως ε, έχουμε χάσει πλέον από τα μάτια μας το στόχο. Και όταν επικρατεί ανασφάλεια απομακρυνόμαστε ο κόσμος απομακρύνεται από το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης και δεν υποβάλλει πλέον αιτήσει. Τις εμπειρίες έχουμε και μάλιστα πάρα πολλέ όταν οι αιτούντες πλέον δεν εστιάζουν στο στόχο αλλά στο πιο εύκολο, αυτό που μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα και πιο ασφαλώς. Αυτό στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και ταχθήκαμε υπέρ μια προσέγγισης την οποία ονομάζουμε Ella Reset Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα τώρα. Από το υφιστάμενο σύστημα, την εικόνα την είδατε και πριν, επιδιώκουμε μια δραστική μείωση των υφιστάμενων συστημάτων. Θέλουμε να απλοποιήσουμε την διοίκηση, τους κανονισμούς, λιγότερες κεντρικές προδιαγραφές, σαφείς κανόνες, λίγες κατευθυντήριες γραμμές και όταν τις έχουμε ως περιγραφή της διαδικασίας και όχι ως νομική προδιαγραφή. Θέλουμε αναλογικότητα. Όλα αυτά θύχθηκαν και από τους προλαλήσαντες. Και φυσικά και εμάς μας απασχολεί το θέμα της εμπιστοσύνης. Φυσικά και χρειάζεται η εμπιστοσύνη σε ένα ελεγκτικό σύστημα το οποίο στο τέλος πρέπει να ελέγχεται και να πιστοποιείται σαφώς και όταν διαπιστώνονται σφάλματα, όταν τα ελεγκτικά συστήματα ελέγχονται και διαπιστώνονται σφάλματα, τότε πρέπει να υλοποιούνται επίσης περαιτέρω έλεγχοι και να επιβάλλονται κυρώσεις. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Στο παράδειγμα που αναφέρατε, κυρία Πρόεδρε, το ελεύθερο κράτος της Αξονίας δήλωσε 2,7% σφαλμάτων ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε 4,4%. Αλλά το ζήτημα είναι πρόκειται για απάτη ή πρόκειται για διαδικαστικά λάθη, παρότι επιτεύχθηκε ο στόχος. Και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή διαφοροποίηση. Και γι' αυτό η προσέγγιση μας έγκυται σε μια σύσπηξη του νομικού πλαισίου, σε έναν προσανατολισμό προς το στόχο και όχι σε μια αιμονή διαδικασία. Και αυτό που ήδη θίξαμε, τον ενιαίο έλεγχο και σαφείς αρμοδιότητες ελέγχου για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να τονίσω μία φορά ακόμα πως είναι σημαντικό για μας. Οι έλεγχοι να αποκαλύπτουν περιπτώσεις απάτης, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να επινηχανέται η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και ο προσανατολισμός προς το στάχο στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποδοχή στο επόμενο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο επειδή δεν είναι δυνατόν Γι' αυτόν τον λόγο επιλέξαμε τον δρόμο να επικοινωνήσουμε σε πολλά κράτη-μέλη για να συζητήσουμε για τις προτάσεις μας με θετικά αποτελέσματα. Δεν είναι δυνατόν. Ακριβώς αυτές οι περιφέρειες για τις οποίες αυτή η χρηματοδότηση είναι πλέον σημαντική να μην μπορεί να την χρησιμοποιήσει. Χρειαζόμαστε μια ριζική επανεκκίνηση. Αυτή, γι' αυτό και αυτή η πρότασή μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία μου εδώ. Ευχαριστούμε και εμείς για κάποιες από τις καινοτόμες προτάσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε σε λίγο. Επειδή ο εσθονός ομιλητής που προβλεπόταν να συμμετάσχει στην ημερήσια διάταξη αναγκάστηκε να μην συμμετάσχει λόγω κυβερνητική κρίση, Δεν θέλει από την πλευρά των κρατών μέλων να κάνει το λόγο η κυρία Περέιρα από την Πορτογαλία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την οργάνωση αυτής της ε, συνάντησης, μια και κάνουμε ένα βήμα προς τα ευρώς προσπαθώντας να βελτιώσουμε ε, τις επιδόσεις μας ε, σε επίπεδο ελέγχων. Η Πορτογαλία θεωρεί πως τέτοιου είδους βελτίωση για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κοινωνιδηλίων είναι απαραίτητη και η ΚΑΠ σίγουρα χρειάζεται κάτι αντίστοιχο. Ξέρετε και εσείς πως είναι από τα κράτη-μέλη που λιγότερο έχουν ωφεληθεί από την κάψη επίπεδο στήριξης της γεωργικής ε, ε παραγωγής και τουλάχιστον σε επίπεδο πρώτου πυλών έχουμε από τη χαμηλότερη επίπεδα στήριξης των ε, εισοδημάτων των γεωργών. Άρα λοιπόν σε οικονομικό επίπεδο η Πορτογαλία βεβαίως έχει ευνοηθεί, ε, ίσως όχι όσο άλλοι. Και αυτό φαίνεται από τα όσα έχουμε επιτύχει και με την άμεση στήριξη και με την έμεση στήριξη όπως επίσης και με τις προσπάθειες προώθησης. Να σας πω πως τα τελευταία 30 χρόνια Εάν δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτή στήριξη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα είχαμε πια αυτό το τόσο σφριγγυλό γεωργικό κλάδο που έχουμε σήμερα στη χώρα μα. Και πρέπει να σα πω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με το επίπεδο στήριξη που έχουμε προσφέρει και εμεί και σε εθνικό επίπεδο. Πάντα είχαμε προβλήματα με την εφαρμογή ε, και την ε, ε, χρήση αυτών των ε, κονδυλίων. Πολλές φορές το πρόβλημα ήταν η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ε, κάποια έλλειψη ευελιξίας στο πώς πρέπει να γίνονται όλες αυτές τις προσπάθειες. Το 2008, για παράδειγμα, μας επιβλήθηκε μια αρκετά μεγάλη διόρθωση γιατί είχαμε προβλήματα με τα συστήματα ελέγχου. Ε, θα πρέπει όμως να δούμε καταρχήν ποιες είναι οι δαπάνες οι οποίες ε, ε, δεν θα έπρεπε να αναγνωρίζονται από τα συστήματα ελέγχου και τα οποία θα έπρεπε να επιστρέφονται αργότερα και να σας πω πως οι έλεγχοι που γίνονται αυτή τη στιγμή οδηγούν σε ανακτήσεις οι οποίες γίνονται με έναν τρόπο που δεν είναι απόλυτα σαφές για τις εθνικές αρχές. Το 2015 πρέπει να σας πω πως οι επιδόσεις μας ήταν κάπως καλύτερες, Πορτογαλία χρηματοδοτήθηκε ε, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και μετά χρειάστηκε να επιστρέψει ένα 3,6% των κονδυλίων που είχε λάβει. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν πως αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ίσως η λύση είναι να βρούμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ τοπικών αρχών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να αποφευθούν τέτοιου είδους ε, προβλήματα στο μέλλον. Να σας μιλήσω για το πρασίνισμα είχαμε πάρα πολλέ αμφιβολίε για το πώ θα πρέπει να ερμηνευθούν οι σχετικέ διατάξει και παρόλε που έχουν γίνει πάρα πολλέ αλλαγέ από τι αρχικές προτάσει, εξακολουθεί αυτό να μένει εξαιρετικά θεωρητικό και να μην είναι ε, εύκολο να εφαρμοστεί επιτόπου από του γεωργού. Θα έπρεπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πρότυπα αυτά να εφαρμόζει μια μεγαλύτερη ευελιξία, παρόλα αυτά θα πρέπει να παραμένουν στη θέση του αυτοί οι στόχοι για το πρασίνισμα, γιατί αν κανεί είναι ε, πολύ αυστηρός τελικά Ειδικά ε, η παραγωγικότητα των γεωργών θα μειωθεί και θα ήθελα να σας δώσω και ένα παράδειγμα Έχουμε κάποιους κανόνες για την ποιότητα των τροφίμων και οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά για τις παραδοσιακές τεχνικές δεν είναι αρκετά ευέλικτες γιατί με τον τρόπο που εκφράζονται δεν μπορούν να Οι παραγωγικοί τρόποι λοιπόν δεν μπορούν να συνεχίζουν να υπάρχουν γιατί κάποιες γαστρονομικές μας παραγωγές και παραδόσεις κόντρεψαν να χαθούν επειδή οι εθνικές αρχές εφάρμοσαν το σύστημα ε, το δικό σας χωρίς καμία ευελιξία. Και η διαφοροποίηση που γίνεται στην Πορτογαλία μεταξύ παραδοσιακών ε, προϊόντων και λοιπών προϊόντων είναι ένας τρόπος για να διατηρήσουμε αυτά τα πάνω από 100 παραδοσιακά προϊόντα που έχουμε ε, στην Πορτογαλία που είναι pop για παράδειγμα ή προστατευμένη γεωγραφική ένδειξη ε, και τα οποία επαναλαμβάνω θέλουμε να διατηρήσουμε και στο μέλλον. Θέλουμε λοιπόν περισσότερο ευέλικτους κανόνες για να μας βοηθήσετε και σε αυτό το θέμα. Καλύτερη, καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές αρχές, περισσότερη ενημέρωση και θα πρέπει ε, να έχουμε και ένα στοχευμένο ε, ε, προϋπολογισμό που θα λάβει υπόψη τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας γιατί είναι τελείως διαφορετική η πραγματικότητα που βιώνουμε, είναι τελείως διαφορετικά τα μοντέλα παραγωγής από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και χρειάζεται να γίνει μια σειρά από προσαρμογέ που θα λάβει υπόψη όλα αυτά τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα και εγώ να πω κάποιους, αναφέρω κάποιου αριθμούς για την ΙΦΑΠ, τον Οργανισμό Πληρωμής στην Πορτογαλία, στην Γεωργική Ανάπτυξη το 2015-2015 αναφέρθηκε ποσοστό σφάλματο 3,3%. Άρα δηλαδή ε, χρήματα τα οποία διατέθηκαν χωρί ε, ε, καμία αιτιολογία, η Κομισιόν είχε αυξήσει το ποσοστό και το 2013 ο ίδιο οργανισμό πληρωμής ανέφερε 2,82% και η Κομισιόν ε, το διόρθωσε, πήγε περίπου στο 4,37 στις άμεσες ενισχύσεις. Ε, φέτος ε, τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Άρα δηλαδή που θέλω να καταλήξω, ότι όταν μιλάμε για απλούστευση θα πρέπει να συζητάμε και για τις, τη μέχρι τώρα απόδοση των οργανισμών ε, πληρωμών. Το λέω αυτό γιατί όλοι μιλήσατε για λιγότερου ελέγχου. Αλλά αφού το λέτε, θα έπρεπε κανεί να μπορεί να εμπιστεύεται περισσότερο του ελέγχου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κουβεντιάσουμε και μεταξύ μα και με την Κομισιόν. Να δούμε πώ θα το καταφέρουμε. Είπατε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών επιτόπου και με εμά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλαούρα από την Ελλάδα και θα ήθελα επίσης ε, να σας πω ότι όσον αφορά τον ελληνικό οργανισμό πληρωμών, ε, πραγματικά ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτόν. Πήγαμε δυο φορές επί τόπου και όσον αφορά την ε, γεωργική ανάπτυξη, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως θα τα θέλαμε. Είπε ο ΠΚΕΠ 2,6 περίπου η Κομισιόν όμως λέει 5,1 ποσοστό σφάλματος. Σας τα λέω έτσι κάπως τους αριθμούς γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί ακριβώς πράγμα συζητάμε έτσι ώστε να μην ε, λέμε διαφορετικά πράγματα. Παρακαλώ κύριε Μπαλαούρα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ε, δεν θέλω να σχολιάσω αναλυτικά τα, τις διαφορές που εντοπίστηκαν ε, διότι όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι ε, υπάρχουν ε, άλλες έρευνες και αναλυτικές καταστάσεις μεταξύ της, του κέντρου, δηλαδή των Βρυξελών και των εθνικών κρατών. Εγώ θέλω να περισσότερο, αλλά αν πάρουμε τα, τα δεδομένα συνολικά, παρατηρούμε, το είπατε και εσείς στην έναρξη της συζήτησης, ότι η μορφή διαχείρισης έχει περιορισμένο αντίκτυπο στο επίπεδο σφάλματος. Το επίπεδο σφάλματος ε, είναι σχεδόν το ίδιο και στους τομείς υποεπιμερισμένη διαχείριση επιτροπής ε, με τα κράτη, μέλη, αλλά και ταυτόχρονα <laughs> στο ίδιο επίπεδο περίπου με δαπάνες από την άμεση διαχείριση της Επιτροπής. Επομένως ε, πρέπει, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, να απλοποιήσουμε ε, και την πολυπλοκότητα που υπάρχει σήμερα και τη γραφειοκρατία ε, έτσι ώστε ο στόχος είναι ε, για να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο είναι απαραίτητος για να εξαλείψουμε και αυτές τις μικρές ε, περιπτώσεις ε, λαθών. Τώρα με αφορμή την συζήτηση που κάνουμε θα ήθελα να, να πω ότι η, θέση μας είναι ότι το σύστημα επιμερισμένης διαχείρισης ε, μεταξύ κρατών και ε, Βρυξελών ε, συμβάλλει, συμβάλλει στην συνυπευθυνότητα και στη συλλογική συμμετοχή ε, στο ευρωπαϊκό όραμα. Η επιμερισμένη ευθύνη αποτελεί ουσιαστική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα πρέπει να διατηρηθεί στο μέλλον αντιμετωπίζοντας ωστόσο την ανάγκη για περαιτέρω απλοποίηση, αναλογικότητα και ευελιξία. Τέλος θα ήθελα να πω, ε, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ότι με την ΚΑΠ, μια και μπήκε αυτό το θέμα, ωφελήθηκαν κυρίως, αν το δει κανένα σε μια ε, χρονική σειρά ε, από την έναρξή της μέχρι σήμερα, πράγματι συνολικά υπήρξε ωφέλεια. Όμως αν ζυγιάσουμε τα κράτη-μέλη θα δούμε ότι τα μεγάλα κράτη εφολήθηκαν πάρα πολύ περισσότερο. Τα μικρά εφολήθηκαν πολύ λιγότερο, αλλά κυρίως δεν υπήρξε πρόνοια για να κατανοήσουν ε, οι Βρυξέλλες ότι, ότι υπάρχουν παραδοσιακές καλλιέργειες και μικροί κλήροι που έπρεπε να τους συντηρήσουν. Επομένως, στα μικρά κράτη δώσαν επιδοτήσεις με συνέπεια οι, οι καλλιεργητές, οι αγρότες να βολεύονται με κάποιες προσωρινές επιδοτήσεις, δεν, αυτό δεν μπορούσε να διακέσει για πάντα, με συνέπεια ας να χαθούν ε, με καλλιέργειες τοπικές που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν ε, την Ευρώπη αφενός και αφετέρου ε, εμείς σαν παράδειγμα στην Ελλάδα ενώ είχαμε συντριπτικό ποσοστό κάλυψη των αγροτικών και κτηνοτροφικών αναγκών μας Τώρα έχει αντιστραφεί τελείω το ποσοστό και μιλάμε για νούμερα 75% αγροτικό τομέα με έναν ήλιο ε, και με ένα ε, κλίμα ε, απίθανο στην Ελλάδα να είναι εισαγόμενο από Ολλανδία, από Γερμανία, από κράτη τα οποία δεν έχουν αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες. Επομένως κάπου υπάρχει το λάθος, εγώ είπα τη γνώμη μου, αν θέλετε το κουβεντιάζουμε αναλυτικά και τέλος θέλω να πω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ακόμα και ευελιξία, δεν είναι το αντικείμενο τόσο της Επιτροπής αυτής, αλλά το, το θέτω για προβληματισμό. Να υπάρχει μια ευελιξία ώστε να βλέπουμε κράτη μικρά που, ε, που μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε εν συνόλο σαν περιφέρειες. Αλλά ακόμα και σαν περιφέρειες να δούμε τι, περιφέρειες των κρατών αυτών, ο οποίος είναι, δεν είναι το ίδιο μια περιφέρεια η οποία είναι σε ε, τριτεύουσα μοίρα σε ένα ε, πλούσιο κράτος με ένα ε, με μια περιφέρεια πολύ φτωχή που είναι σε ένα φτωχό κράτο και έχει σε ένα κράτο με κρίση. Άρα ε, πρέπει και η, Επιτροπή μα να, να δώσει έμφαση και να επαναφέρει την, ε, τη, τη, τη, συνθήκη, το άρθρο της συνθήκης για τη σύγκληση, γιατί τώρα που ήταν αγοργωνιαίος λήθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τώρα βλέπουμε συνεχώς αποκλήσεις. Συνεχώ αποκλείσει σε όλα τα δεδομένα, όχι μόνο στον αγροτικό τομέα ή στα άλλα περιφερειακά ε, δρόμενα, αλλά έχουμε αποκλησει Ας πω ένα παράδειγμα, η Γερμανία έχει πλεόνασμα στο δημοσιονομικά τη, έχει 9% του ΑΕΠ. Όταν αυτό απογορεύεται από τι συνθήκε. και όταν ένα κράτο τολμήσει να έχει έλλειμμα πάνω από τι συνθήκε, τότε του πιάνουν το αυτοί και του τιμωρούν. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα συζητήσουμε κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τον συνάδελφο κ. Μαρτίνη από τη Γερουσία της Ιταλίας. Τώρα πάλι θα αναφερθώ σε αριθμούς στην αγροτική ανάπτυξη. Υπάρχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα τα οποία έχουν βελτιωθεί στην Ιταλία αλλά μας έχει δηλωθεί μια τιμή 1,35% η οποία διορθώθηκε σε 5,12%. Αλλά οι άμεσες ενισχύσεις είναι πολύ σημαντικές επειδή εκεί καταβάλλονται μεγάλα ποσά και εκεί μόνο μία τιμή βρίσκεται πάνω από το όριο του 2%. αλλά πιστεύω πως από κοινού θα ήμασταν ισχυρότεροι αν ενώναμε τις δυνάμεις μας. Κύριε Μαρτίνη. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένους αριθμούς, ούτε θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες πολιτικές, αλλά θέλω να σας πω ότι ήρθα εδώ για να σας πω ότι η Ιταλική Γερουσία ε, τάσεται υπέρ του να ελέγχεται ο προϋπολογισμός και αυτό να κρυθεί ως ένα μόνιμο σύστημα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα και για να μπορέσουμε από κοινού να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρό. Ω Ως γερουσία θέλω να σας πω ότι καταφέραμε πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Από το 2009 είχαμε μία αρχική έρευνα σχετικά με τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων και του συναφείς ελέγχους και κάναμε, υποβάλαμε προτάσεις ε, στην κυβέρνηση με βάση αυτή την ανάλυση, γιατί είχαν αποκαλυφθεί και ελλείψεις ε, σε επίπεδο διαχείρισης, γραφειοκρατίας. Είχε αποδειχθεί ότι υπήρχαν και ελλείψεις στους εκτονιστέρων των ελέγχους. Αυτή λοιπόν όλη η δουλειά απέδωσε και όπως αναφέρθηκε πράγματι υπάρχει κάποια βελτίωση ε, το σύστημα της Μαρτίους, του Μαρτίου κατέδειξε ότι έχουμε ε, κονδύλια που ε, ε, επιδεικνύουν μια σημαντική απορροφητικότητα. Αυτό για την Ιταλία είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η κυβέρνηση έχει ορίσει μια, ένα συγκεκριμένο οργανισμό ο οποίος καταλήγει στα συμπεράσματα και υπάρχουν περιφέρειες ε, οι οποίες έχουν κινητοποιηθεί. Εμείς λοιπόν δώσαμε κίνητρα για να σκέφτονται όλοι αυτοί οι οργανισμοί με ευρωπαϊκά κριτήρια. Εγώ πριν γίνω γερουσιαστής ήμουνα περιφερειάρχη στην Τοσκάνη για 10 περίπου χρόνια Φαντάζομαι ειδικά οι Γερμανοί φίλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την περιοχή μα. Και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω μια συζήτηση που γινόταν τότε στην Επιτροπή των Περιφερειών. Λέγαμε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν ήταν να περιφερειοποιηθεί η Ευρώπη, αντίθετα να εξευρωπαϊστούν οι περιφέρειες, δηλαδή να χρησιμοποιούνται σωστά τα κονδύλια που υπάρχουν για την εφαρμογή ευρωπαϊκή πολιτική. Τελειώνοντα, θέλω να σα πω ότι η δική μα η Γερουσία στι 22 Νοεμβρίου ε, θα ε, φιλοξενήσει ένα σχετικό σεμινάριο όπου θα παρουσιαστεί η ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Και αυτή είναι μία μορφή συνεργασίας. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι εμείς ελπίζουμε να μπορέσουμε να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, να βελτιωθούν τα στοιχεία για να υπάρχει καλύτερη ε, ταυτοποίηση και ταύτιση μάλλον των στοιχείων που δίνει η ε, δική μας η κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι να εντοπιστούν ε, βέλτιστες πρακτικές για, το χρήσο, το, για τη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Βεβαίως ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και να ξεπεράσουμε αυτή την αρχή use it or lose it, αλλά ξέρω ότι αργότερα υπάρχει μια ειδική συνεδρία που θα εξετάσει το θέμα αυτό, άρα δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Είναι όμως χρήσιμο και σημαντικό αυτό το εργαλείο για να βοηθηθούν οι περιφέρειες. Τελειώνοντας και πάλι θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχουν μορφές συνεργασίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, κυρίως με την Επιτροπή για τον Έλεγχο των Προπολογισμών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Τα θέματα αυτά δεν είναι δημοφιλή στα κράτη-μέλη, πρέπει να το πούμε αυτό. Γνωρίζουμε πως τα κράτη-μέλη διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο όσον αφορά τον χειρισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής, έχουν διαφορετικούς διοικητικούς οργανισμούς και έχουμε κράτη-μέλη με πολλά ή λιγότερα προβλήματα και θα επιθυμούσαμε τα εθνικά κοινοβούλια κυρίως των χωρών αυτών που έχουν περισσότερα προβλήματα να επιλαμβάνονται περισσότερο των θεμάτων αυτών. Δεν αποτελεί μυστικό. Η Ιταλία είναι μία από τις χώρες, όπως και η Ισπανία, με μία από τις χώρες με τα περισσότερα προβλήματα και μπορούν να ξοδευτούν τεράστια ποσά χρημάτων και καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες να επιτύχουμε καλά αποτελέσματα στην Ελλάδα και στην Επιτροπή αυτή χτες ε, θίξαμε τα διαθρωτικά προγράμματα. Με πολύ καλή βούληση προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Στα γεωρικά ταμεία, θα δώσω στον κύριο Μέβελε πάλι το λόγο, και έχουμε το πρόβλημα ότι έχουμε 100% Έλέγχο στα χαρτιά, αλλά επιτόπου ο έλεγχο αναρχείται στο 5% ή και λιγότερο. Και σε αυτούς σε αυτό το 5% των περιπτώσεων ο έλεγχος είναι πολύ έντονος. Φυσικά και βρισκόμαστε επί τόπου επειδή πρέπει να δικαιολογήσουμε τα χρήματα των φορολογουμένων. Απλά το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα το σύστημα αυτό. Πρόκειται για ένα συστημικό ερώτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε πιο έντονα. Οπότε παρατηρούμε το πρόβλημα από τη μία και από την άλλη πλευρά και φτάνουμε στο συμπέρασμα πω πρόκειται για ένα σύστημα που είναι ακόμα λιγότερο γραφειοκρατικό. Είμαι εδώ και 13 χρόνια μέλο τη επιτροπή και λυπούμε. Δεν έχω κάποια καλύτερη ιδέα. Εάν έχετε κάποια καλύτερη ιδέα πείτε την. Αλλά εμεί, επί του παρόντο, βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσχερή θέση επειδή φυσικά και βλέπουμε σαφώ συγκεκριμένα προβλήματα στα κράτη-μέλη, αλλά δεν έχουμε λύσει. Οπότε ο κύριο Μέβελε πρέπει να μα μιλήσει για τι λύσει. Κύριε Μέβελε. Ευχαριστώ πολύ. Nothing, nothing easier. Το πιο εύκολο είναι αυτό που μου ζητάτε. Να ξεκινήσω λοιπόν με την τελευταία σας παρατήρηση, γιατί νομίζω ότι φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα ελέγχων, με τον τρόπο που αυτοί διεκπαιρώνται τώρα. Μιλήσατε για 100% διοικητικού ελέγχου και μόνο 5% επιτοπίου ελέγχου. Βεβαίω ποτέ δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο 5% επιτοπίου αν δεν είχαμε τη δυνατότητα του 100% διοικητικού ελέγχου που πρέπει να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά λεπτομερείς και κυρίως για το μεγάλο βαθμό ε, των ε, ελέγχων που γίνονται για, τους, ε, για τις εκτατικές επιδοτήσεις. Και ό,τι γίνεται στα πλαίσια του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχαίων, να σας πω πως το εργαλείο αυτό λειτουργεί πολύ σωστά στα χέρια πολλών κρατών μελών. Και θα επανέλθω τώρα στις δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά για το θέμα του LPIS. Έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Για την Πορτογαλία να σας πω ότι ότι ο κύριος Περέιρα από την Βουλή της Πορτογαλίας μίλησε για τους καταλογισμούς του 2008 και ε, μετά που σχετιζόντουσαν πάντα σε προβλήματα που υπήρχαν με τα μέτρα τα εκτατικά, γιατί το σύστημα αναγνώριση αγροτεμαχίων δεν ήταν ενημερωμένο και πάρα πολλέ μη επιλέξιμε εκτέσει είχαν τοποθετηθεί το σύστημα. Όλα αυτά έχουν ξεκαθαρίσει και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συγχαρώ τον Οργανισμό Πληρωμών τη Πορτογαλία γιατί το έκανε. Ήταν πολλέ οι προσπάθειε που έγιναν, πολύ δύσκολη η διαδικασία, αλλά νομίζω ότι εκεί σημειώσαν πάρα πολύ πρόοδο. Μία αντίστοιχη δήλωση που να κάνω και για την Ελλάδα. Γιατί και εκεί, εδώ και χρόνια συνεργαζόμαστε με τους Έλληνες συναδέλφους και έχουμε πάει θαυμάσια. Νομίζω ότι μπορώ να πω πια ότι το σύστημα λειτουργεί και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να καλέσω την ελληνική, το ελληνικό κοινοβούλιο να εξασφαλίσει πως το σύστημα θα συντηρηθεί και θα ενημερώνεται σε τακτικά διαστήματα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε πως αυτή η έπαινη που εκφράζω θα συνεχίσουν να ακούγονται και σε δύο-τρία χρόνια και δεν θα είναι ε, έπαινοι μόνο για τη συγκεκριμένη χρονιά. Βεβαίως υπάρχει πολύ πρόοδος και όταν καταλήγει σε ένα 2,9 ε, ποσοστό σφάλματος για τον πρώτο πυλόν ε, και δύο, δεύτερο πυλόν και 2,2 για τον πρώτο πυλόν, τα πράγματα είναι, πάνε καλά. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για όλους και έχουμε ακόμα οργανισμούς πληρωμών όπου χρειάζεται πολύ προσπάθεια και Έχουμε και πάρα πολλές υποθέσεις και περιπτώσεις όπου τα πράγματα λειτουργούν πολύ καλύτερα, χάρη όμως κυρίως στα συστήματα και κυρίως στον ΩΣΔΕ που ενημερώνονται ε, κατάλληλα, έτσι ώστε να λειτουργούν σωστά. Θέλω να πω και κάποια ε, λόγια ακόμα, ξεκινώντας από τα όσα είπε ο Υπουργός κ. Σμιτ. Πρέπει να σας πω ότι αυτά που είπε τα πήχησαν και άλλοι και έκανε μια διάκριση μεταξύ απάτης και τυπικών σφαλμάτων. Ε, εγώ είμαι ένα αξιωματούχο που προετοιμάζει την απαλλαγή για τον Επιτροπό μου και πρέπει να σα πω πω θα πρέπει να βασίζομαι στι νομικέ διατάξει, οι οποίε οι ίδιε δεν κάνουν αυτή τη διάκριση μεταξύ σφαλμάτων και δεν μιλά για κάτι τέτοιο, μιλά για νομιμότητα και κανονικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε όλες τις συναλλαγές οι οποίες δεν γίνονται ευθυγραμμισμένα με τις νομικές διατάξεις και που οδηγούν σε πληρωμές οι οποίες είναι αχρεωστήτως καταβληθήσεις. Και αν εμπλέκεται βεβαίω, αν υπάρχει και διάσταση απάτης, τότε ναι, θα πρέπει η εισαγγελία και οι εθνικές αρχές να πατάξουν αυτή την απάτη. Αν όμως μιλάμε ε, για θέματα τα οποία ε, χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό, ε, κοιτάξτε, το μόνο συμπέρασμα είναι ότι οι κανόνε είναι πάρα πολύ σαφείς. Ναι, ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτεί αυτές τις ε, προσπάθειες. Τώρα, για τις νομικέ διατάξει, στις οποίε αναφερθήκατε δεν ξέρω αν η, προ... η πρόταση που προβάλλεται είναι μία την οποία θα θέλαμε να την ε, δεχτούμε και Τώρα για το θέμα της απάτης, άκουσα ότι είπε ο πρόεδρος Καλντέρα όταν παρουσίασε την ετήσια έκθεση, δεν είναι το πρόβλημα η απάτη σήμερα. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα συστήματα ελέγχου δεν λειτουργούν σωστά. Και έτσι έχουμε μη επιλέξιμες ε, εκτάσεις που καταχωρούνται, για παράδειγμα, προθεσμίες που δεν γίνονται σεβαστέ τέτοιου είδους προβλήματα. Και δεν μπορούμε απλώς να αμελήσουμε αυτού του είδου τα σφάλματα, αλλά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να εξασφαλίσουμε πως δεν θα συμβαίνουν. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση αυτή που γίνεται. Επίση, δέχομαι πως το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο απλό, έτσι ώστε να μην έχουμε καταλογισμούς. Ε, και νομίζω ότι ποτέ δεν είναι ευχάριστο να έχει κανεί μια τέτοιου είδου οικονομική διόρθωση, γιατί πετά χρειάζεται κανεί τον προπολογισμό να βρει τα κονδύλια για αυτήν. Όμω δεν θα πρέπει να υπερεκτιμήσουμε το μέγεθο του προβλήματο, γιατί αυτοί οι καταλογισμοί, του οποίου κάνει η Γενική μου Διεύθυνση κάθε χρόνο, είναι γύρω στο 2% τη ε, συνολική δαπάνη για την ΚΑΠ. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ποσοστό που του είναι σχετικά μετρημένο και αυτό σχετίζεται και με τη δήλωση που έκανα πως η κατάσταση στους οργανισμούς πληρωμών δεν είναι η ίδια παντού. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου οι καταλογισμοί είναι υψηλότεροι και υπάρχουν κράτη-μέλη όπου είναι χαμηλότεροι. Τώρα, δεν θα κατονομάσω κράτη-μέλη, ούτε αυτούς που έχουν πάει καλά, ούτε αυτούς που έχουν πάει άσχημα, όμως στο παρελθόν πρέπει να σας πω ότι έχουμε αντιμετωπίσει ε, πρόβλημα όπου σε περιπτώσεις που είχαμε χαμηλούς καταλογισμούς οι αντιδράσεις ήταν εξαιρετικά ε, θορυβώδεις. Άρα λοιπόν το να λειτουργούν τα πράγματα σωστά ε, ουσιαστικά οδηγεί κάποιους να πιστεύουν πως στα δικά μου χωράφια εμείς ε, λάθη δεν κάνουμε και πολλές φορές για μικρό καταλογισμό να ακούσει κανείς πολλές αντιδράσεις. Αλλά όταν έχεις ένα μεγάλο προπολογισμό πολύ συχνά μπορεί να κάνεις κάποιο λάθος και ένα τέτοιο σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε μια οικονομική διόρθωση. Μιλήσατε και για τις κατευθυντήριες γραμμές και μας είπατε πως είναι υπερβολικές. Ναι, αλλά αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές συνήθως ε, συγγράφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν ετήματος των κρατών μελών. Γιατί τα κράτη-μέλη θεωρούν πως το νομικό πλαίσιο αφήνει παραθυράκια ανοιχτά, τα οποία χρειάζεται να γίνουν πιο συγκεκριμένα και ή να αποφευθούν αργότερα οι καταλογισμοί, τα κράτη-μέλη και οι οργανισμοί πληροφών πολλές φορές θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το σκεπτικό της Κομισιόν για κάποιες νομικές διατάξεις, οι οποίες ενδεχομένως δεν είναι αρκετά σαφείς ή είναι κάπως γενικόλογες. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας ε, αδυσόπιτος κύκλος όπου αφενός μας ζητάνε να δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολισμούς και όταν το κάνουμε και δεν γίνονται σεβαστές τότε να πούμε «Α, εντάξει δεν πειράζει γιατί στο κάτω-κάτω κατευθυντήριες γραμμές ήταν, δεν ήταν δεσμευτικές». Ε, άρα λοιπόν ε, να μην ε, προσπαθούμε μετά να διορθωθούν όλα αυτά μέσω ε, καταλογισμών. Είναι ένα δίλημα το οποίο δεν βλέπω έναν εύκολο τρόπο να ξεπεράσουμε παρά μόνο τα όσα πρότεινα στην παρουσίασή μου και νομίζω πως η απλούστευση είναι ένας από τους τρόπους να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Γιατί έχουμε το εφαρμοστικό πλαίσιο μεν, αλλά θα πρέπει να δούμε και τους ουσιαστικού κανόνες στους οποίους προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Γιατί αν καταφέρουμε ε, να αποκλιμακώσουμε την, το πόσο περίπλοκο, περίπλοκη είναι αυτή η, η νομοθεσία, η έλεγχη θα γίνει πιο απλή και λιγότερο επιβαρυντική. Κύριε Περέιρα, μιλήσατε για το πρασίνισμα, που είναι υπερβολικά θεωρητικό ή περίπλοκο έτσι όπως περιγράφεται. Αυτό αποφασίστηκε πριν από δύο-τρία χρόνια. Και ξέρετε πως το έχουμε εφαρμόσει, νομίζω, είναι η πρώτη φορά ή η δεύτερη φορά το 2016. Ο Επίτροπός μου ε, μόλις πρότεινε μια σειρά απλουστεύσεων για το πρασίνισμα και βεβαίως αυτό θα αποτελέσει και ένα θέμα μεγάλης συζήτησης και σε επίπεδο κοινή γνώμης αλλά και σε επίπεδο ε, ελεγκτικού συνεδρίου το οποίο μόλις ξεκίνησε να συγγράφει μια ε, συγκεκριμένη έκθεση για το σύστημα του περσινίσματος και στα, στα φώτα των όσων περιγράφει αυτή η έκθεση θα δούμε αν το σύστημα θα συνεχίσει να υφίσταται ως έχει ή αν θα κάνουμε κάποιες ουσιαστικές τροποποίησεις. Κατανοώ επίσης την ανάγκη για ευελιξία και θα ήθελα να σας καλέσω όμως όλους ζητάνε ευελιξία να μου εξηγήσουν ακριβώς τι σημαίνει. Ο κύριος Περέρα αναφέρθηκε στις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και στα ΠΟΠ και στο ότι δεν είναι αρκετά ε, ευελικτά αυτά τα σχήματα. Συγγνώμη, 200 τέτοιες παραδοσιανεμικές ονομασίες έχετε στην Πορτογαλία. Άρα δεν μπορεί να είναι και πολύ δύσκολο να το πετύχει κανεί. Και να σα πω πω τέλο θα πρέπει να δεχτούμε πω μιλάμε για δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, τα οποία χρειάζεται να πλαισιώνονται και να περιγράφονται με ένα σαφή και ενδεχομένω και λίγο αυστηρό τρόπο καμιά φορά έτσι ώστε να εφαρμόζονται και επιτόπου, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την κατάχρηση αυτών των ονομασιών από όσους δεν σέβονται τις προϋποθέσεις για την απόκτηση αυτής της ονομασίας. Μια τελευταία παρατήρηση για το θέμα της απλούστευσης. Σκεφτόμουν το θέμα και κατέληξα στο ότι η μεγάλη αλλαγή στην ΚΑΠ και η οποία ενεργοποίησε όλα αυτά τα ε, παράπονα για του πόσο περίπλοκα είναι όλα αυτά. Ε, όλα αυτά συνέβησαν το 1992 όταν φύγαμε από μια πολιτική αγορά σε μια πολιτική στήριξη εισοδήματο. Μετά από αυτό βεβαίω είχαμε την μεταρρύθμιση Φίσλερ το 2003 και μετά εφαρμόσαμε ένα σύστημα που είναι στήριξη εισοδήματο. Πριν το 1992 η παραγωγή δεν ήταν τόσο ενταγμένοι στο σύστημα. Έφερναν, το παραγω... Έφερναν τα προϊόντα τους στην παρέμβαση, αποθηκευότανε, ε, ε, γινόταν εξαγωγή, είχαμε μια στήριξη της τιμής από την ευρωπαϊκή κοινότητα όπως ονομαζόταν τότε, αλλά από το 1992 και μετά οι Γεωργοί αποτέλεσαν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ίδιου του συστήματος, δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνονται πληρωμές σε 8 εκατομμύρια ε, γεωργούς στον πρώτο πυλώνα και σε 2,5 στο δεύτερο. Άρα το 5% ε, επιτόπιοι έλεγχοι μιλάμε για περίπου 1 εκατομμύριο ε, επιτοπίους ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. Άρα λοιπόν συζητώντας τα νούμερα αυτά βλέπουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό προτείνατε και εσείς κύριε Σμιτ, κύριε Υπουργέ, και το είπα και εγώ στην αρχική μου δήλωση. Θα πρέπει να μετακινηθούμε από ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ περίπλοκο για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να επαναπροσανατολίσουμε την πολιτική μας σε στόχους, σε απόδοση, σε αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει να επιτυγχάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι αισιόδοξο πως αυτό θα λειτουργήσει. αλλά πρέπει το σύστημα αυτό να το διαμορφώσουμε με έναν τρόπο που δεν θα μα οδηγήσει στα ίδια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα με τη συμμόρφωση, τουλάχιστον όταν τη δούμε από τη σκοπιά τη απόδοση. Δηλαδή, να μην έχουμε στόχους απόδοσης που θα είναι τόσο εξελιγμένοι που θα μπορεί κανείς να τους πετύχει και να τους παρακολουθήσει και να τους εποπτεύσει μέσω ενός εξαιρετικού περίπλοκου σύστημα παρακολούθησης και πλαισίου ε, εφαρμογής. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Νομίζω όμω πω αυτό θα πρέπει να έχουμε κατά νου όταν το συζητάμε, γιατί τώρα βεβαίω είναι το μαγικό ραβδί, στο μέλλον θα έχουμε την αποδοτικότητα και στα επόμενα προγράμματα θα μετράμε δείκτες απόδοση σε σχέση με προκαθορισμένου στόχου κτλ. Αλλά αυτά μπορεί να μα οδηγήσουν, και γι' αυτό το είπα στην αρχική μου δήλωση, να αποφύγουμε τέτοιου είδους ε, ε, διατάξεις σε επίπεδο τελικού δικαιούχου, γιατί τότε οι τελικοί δικαιούχοι θα δυσκολεύονται πάρα πολύ, αλλά να το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο γιατί αν ακολουθήσουμε την ίδια άγουσα που ακολουθήσαμε με την συμμόρφωση, θα δείτε πως θα αντιμετωπίσουμε και για την απόδοση ακριβώς τέτοια προβλήματα στο μέλλον. Βεβαίως, όνειρο είναι αυτό το να παράγει κανείς ό,τι θέλει και ξαφνικά να έρχεται κάποιος και να πληρώνει. Ε, δεν πάει έτσι. Ούτε πρόκειται να λειτουργήσει έτσι. Και στο μέλλον μάλιστα ακόμα λιγότερο επειδή θα υπάρχει ε, πρόβλημα οικονομικό. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λαζάρου από το Ελεκτικό Συνέδριο για να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε στον γεωργικό τομέα γιατί εδώ ξέρετε τι γίνεται ε, κατ' ουσίαν ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, η Κομισιόν ε, απευθύνεται στο λεκτικό Συνέδριο, το λεκτικό Συνέδριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι είδους συζητήσεις γίνονται τώρα στο λεκτικό Συνέδριο, έτσι ώστε αυτό το μαγικό 2% που αναφέρεται, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό, ε, συζητάτε εσείς στο ελεγκτικό συνέδριο, θέλετε να αλλάξετε κάτι ή θα μείνουν όλα όσα έχουν. Ε, κύριε Λαζάρου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Um, indeed, as um, the Commission... Ευχαριστώ, κύριε Επιτροπή. Ε, improvement in, the, in Pillar Wall. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Ε, υπάρχει πράγματι βελτίωση στο ποσοστό σφάλματος ε, στον τομέα της γεωργίας. Και, βεβαίως και υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά. Ε, γνωρίζουμε και σημειώσαμε ότι η συνεισφορά γενικά στο ποσοστό σφάλματος στον τομέα της γεωργίας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, το ποσοστό σφάλματος στον τομέα της γεωργίας παραμένει το ίδιο αν συγκρίνουμε το 14 και το 15. Το γνωρίζουμε αυτό και το διαπιστώσαμε. Γνωρίζουμε όμως επίσης Γνωρίζουμε όμως ότι έχει υπάρξει και βελτίωση στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων. Δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη επαγρύπνηση, κυρίως από πλευράς ε, των ε, δημόσιων αρχών. Επίσης ε, υπάρχει και η προοπτική να μειωθεί το ποσοστό του σφάλματος στην, στον τομέα των άμεσων ενισχύσεων. μας ρωτήσατε τι σκοπεύουμε να κάνουμε εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο. Και όπως σας ανέφερα ήδη, εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση στους ελέγχους και εξετάζουμε τρόπους για το πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τις Εθνικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρουν ε, περισσότερα, περισσότερο ασφαλή στοιχεία συμμόρφωσης έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε να βασιστούμε περισσότερο στη δική τους τη δουλειά, τη δουλειά του ελέγχου. Και να μπορούμε και εμείς να τοποθετούμε στους, ε, στα στοιχεία που μας ε, υποβάλλουν. Εμείς ελπίζουμε μέσα από τη δική μας τη δουλειά, τη δουλειά των ελέγχων, θα ενθαρρύνουμε και την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να ε, συμβάλλουν στο να υπάρχουν περισσότερο αξιόπιστα στοιχεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Σμιτ, ε, πολύ μου άρεσαν αυτά που είπατε με τους αριθμούς, κυρίως σχετικά ε, με τους ε, τρεις κανονισμούς που διαγράφηκαν ο Έζη, παραδείγματος χάρη, που βέβαια δεν άρεσε αυτό σε μερικούς τον προπολισμό, αλλά τι να κάνουμε, μετά ένας άλλος κανονισμός στον γεωργικό τομέα, ούτε και εμένα μου άρεσε αυτό, τι να κάνω, ε, πράγματι όμως πρέπει να δεχτώ ότι απελευθερώνονται νέες δυνατότητες. Αυτό που με απασχολεί λιγάκι είναι το ότι κατ' ουσίαν θα υποφεληθούν εκείνοι οι οποίοι όμως μέχρι τώρα δεν είχαν να επιδείξουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, πώς θα μπορέσουμε να διαβεβαιώσουμε τους φορολογούμενους ότι γίνεται η βέλτιστη χρήση των χρημάτων τους. Στη Βάδη Βιτεμβέργη, εκεί ε, πρέπει κανένα το δει λιγάκι, παραδείγματος χάρη, το, τη στοιχίζει όλο αυτό. Και αυτό που μας απασχολεί είναι πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, να μην υπάρχει το δίλημα. Δηλαδή να υπάρχει και αξιοπιστία, να υπάρχει εκφοβισμός, ε, γιατί εσείς μιλήσατε για το θέμα αυτό του εκφοβισμού, πώς μπορούμε να τα καταργήσουμε όλα αυτά, χωρίς όμως να καταλήξουμε σε ένα σύστημα όπως αυτό που παρουσίασε ο κύριος ε, Μέγκουλε. Να πω πολύ σύντομα στον κύριο Μέγκουλε ότι τον ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν τον βλέπω εδώ για πρώτη φορά και ως εκ τούτου πολλά από αυτά που είπε ε, τα έχω ξανακούσει. Αυτή η single audit προσέγγιση έχει ξαναναφερθεί υπάρχει σχετικό αίτημα. Αυτό που δεν προβλήθηκε πολύ είναι το θέμα της Ευρώπης. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση. Εμείς ε, θέλουμε να καταπολεμηθεί αυτή η απογοήτευση που υπάρχει για ευρωπαϊκά θέματα. Και αυτό το ανέφεραν και πολλοί άλλοι. Εγώ δεν είμαι, δεν ανήκω σε εκείνους που λένε ότι αυτά που σκέπτονται οι Βρυξέλλες είναι ομολόχ της γραφειοκρατίας. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για πολλά πράγματα φταίνε οι περιφέρειες, ε, φταίνουν τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν οι Βρυξέλλες που αποφασίζουν ορισμένα πράγματα, αλλά τι προκύπτει ε, το θέμα δεν είναι ποιο είναι υπέτειο, το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να πλουστεύσει το σύστημα και να στρέψει το βλέμμα προς τα εμπρός. Ε, εγώ θα πω κάτι άλλο, κάτι που έχει σχέση με αυτό που ρωτήσατε εσείς. Δηλαδή, στη Γερμανία τα ΙΧ μέσα από ε, οργανισμούς πιστοποίησης ελέγχονται από τον ΤΟΥΦ, από την ΤΕΚΡΑ και το κράτος τι κάνει, αναθέτει την πιστοποίηση σε ένα συγκεκριμένο αναγνωρισμένο φορέα, ο οποίος ελέγχεται. Ελέγχεται ο φορέας κατά πόσον τηρεί όλες τις ε, προδιαγραφές για να κάνει αυτό το αρκετά να εκτελεί αυτό το περίπλοκο καθήκον. Έτσι λοιπόν κάπως πρέπει να λειτουργεί το όλο σύστημα. Δηλαδή η Ευρώπη, ανάλογα με το που θα βρίσκονται οι αρμόδιες διοικητικές αρχές, η Ευρώπη θα πρέπει να πιστοποιήσει τους οργανισμούς πληρωμής να τους ελέγχει βέβαια και οπουδήποτε προκύπτουν προβλήματα, εκεί θα παρεμβαίνει η Ευρώπη. Δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού, αλλά αν θέλετε να υπάρχει ένα σύστημα όπου εκεί όπου τα πράγματα λειτουργούν εύρυθμα, εκεί όπου υπάρχει εμπιστοσύνη, να μπορεί κανείς να πει εντάξει, εσείς λειτουργείτε μια χαρά, συνεχίζετε. Σίγουρα ο οργανισμός αυτός θα ελέγχεται κατά καιρού, αλλά οποτεδήποτε διαπιστώνει κανείς ότι όλα πάνε μια χαρά, το αυτός απίνεται να λειτουργεί περαιτέρω. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά, εκεί θα πρέπει να δει, τι πρέπει να, να δει τι πρέπει να γίνει με τον οργανισμό πληρωμή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το να κάνουμε αυτό το, σύστημα, να εφαρμόσουμε το σύστημα, να υπάρχει εμπιστοσύνη και στην περίπτωση αυτή, αν γίνουν έτσι τα πράγματα, μπορούμε να περιορίσουμε τους ελέγχους και μπορούμε σε μεμονωμένες περιφέρειες να διεξάγουμε μεμονωμένους ελέγχους ανάλογα με τα αποτελέσματα που υποβάλλονται. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα και που δεν αναφέρθηκε όμως είναι το εξής. Να σκεφτούμε το κατά το θέμα της απλούστευσης της διοίκησης που πολλοί το έπτυξαν, κατά πόσον αυτό μπορούμε να το αποκόψουμε από άλλα αιτήματα. Νομίζω πρέπει να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός. Γιατί τελικά το θέμα δεν είναι κατά πόσον γίνονται χι επενδύσεις στη γεωργία, υπάρχει γεωργική ανάπτυξη. Η διοίκηση εμπλέκεται με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω, ίσως ε, ε, θα μπορούμε παράλληλα να συζητάμε, πάντως όχι σε συνδυασμό. Σίγουρα όχι σε συνδυασμό. Αυτά που συζητάμε με γεωργική ανάπτυξη, παραδείγματος χάρη. Ε, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή πολλά κρατημέλη αντιμετωπίζουν την ε, Ευρώπη με επικριτικό πνεύμα. Ε, όμως, ξέρετε, μια ισχυρή Ευρώπη ποτέ δεν την είχαμε ανάγκη όσο σήμερα. Αν ρίξουμε έτσι μια ματιά στο διεθνές γίγνεσθε. Άρα, δηλαδή, μας ενδιαφέρει να υπάρχει αποδοχή, αποδοχή της Ευρώπης που θα την επιτύχουμε όπως σας ανέφερα. Ευχαριστούμε για την συμβολή σας στην συζήτηση, το σύστημα με μπόνους και με άλλους. Σαν την περασμένη φορά την εισηγήτρια, τα κράτη-μέλη την απέρριψαν, αλλά και πάλι έχουμε την ευκαιρία με αυτή τη μεταρρύθμιση και αυτή την τροπολογία θα την καταθέσουμε και πάλι και θα γίνει γρήγορα, επειδή έχει ήδη συγγραφεί και ήδη έχουμε ανταλλάξει απόψει με τα κράτη-μέλη γι' αυτό και θεωρώ πως είναι πρωτοπόρο αυτό και καλό να λύσουμε επιτέλους τα προβλήματα και που είναι και όχι συνέχεια να τιμωρούμε. Οι παρατηρήσει σα βέβαια βρίσκουν γόνιμο έδαφο σε εμά. Περνούμε στο δεύτερο τμήμα, η ανοησία του use it or lose it προς ένα σύστημα που κινείται περισσότερο από την απόδοση για τα τζαπάνες. Καλωσορίζουμε εδώ. Το λόγο έχει ο κύριος Λαζάρου από το Ελεκτικό Συνέδριο. Thank you, uh, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μιλήσουμε λοιπόν για την αποδοτικότητα ως ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολεί. Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 η είχαμε το use it or lose it, δηλαδή στόχο μας την απορρόφηση και περισσότερο την ε, συμμόρφωση παρά την καλή απόδοση. Δηλαδή τα έργα τα οποία χρηματοδόθηκαν εστίαζαν περισσότερο στην δαπάνη των υφιστάμενων ευρωπαϊκών κονδυλίων, μετά στη συμμόρφωση με τους κανόνες και τέλος και σε περιορισμένο επίπεδο με την επίτευξη των στόχων και των επιπτώσεων. Αυτή η έλλειψη στόχευση των αποδόσεων αποτελεί και ένα από τα βασικά προβλήματα στο σχεδιασμό του ευρωπαϊκού περιπολογισμού αυτό ήταν το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε σε αυτή την, στον ευρωπαϊκό έλεγχο που κάναμε για τα ε, σχετικά θέματα του 2013. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως η Επίτροπος κυρία Γεωργίευα ξεκίνησε μια εκστρατεία να αλλάξει αυτή η νοοτροπία και να γίνει ο προπολογισμό Ευρωπαϊκό, ένας προπολογισμό που εστιάζει στα αποτελέσματα. Του ενθαρρύνουμε. Η απορρόφηση, η δυνατότητα χρήσης των κατανεμημένων κονδυλίων βεβαίως αποτελούν ένα βασικό στοιχείο τη διαχείριση και στην ετήσια έκθεση της, σχετικού τμήματος για την Ευρωπαϊκή Περιοχή, Περιφερειακή ε, πολιτική ακούστηκε ε, πως ε, τα αποτελέσματα της ομάδας δράσης που στήθηκε το 2014 για να αυξήσουν την απορροφικότητά τους στα κράτη που είχαν μικρότερη απορροφικότητα, κατέληξε στο ότι η επιδόση απορροφητικότητας είναι διαφορετική για τα 28 κράτη-μέλη. Σε κάποια κράτη-μέλη είναι μειωμένη η απορροφητικότητα σε σχέση με τη δημόσια δαπάνη. Για άλλα κράτη-μέλη τα ποσά, τα οποία είναι ακόμα προς απορρόφηση είναι ένα βασικό κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων. Στην δική μας έκθεση φέτος ε, συστήσαμε να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δυναμικό, το περιορισμένο δυναμικό κάποιων κρατών μελών έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τα κονδύλια αυτά με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, γίνεται το κυρίαρχο στοιχείο επιλογής έργων σε κάποια κράτη-μέλη και το αποδείξαμε αυτό σε μια ανάλυση που κάναμε σε μια ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου το 2014. Δηλαδή για τα εκολαπτήρια ε, επιχειρηματικότητας τα business incubators είδαμε πως υπάρχει μια δυναμία στα κριτήρια επιλογής και για τις ε, φιλοξενούμενες εταιρείες υπάρχουν γενείς αδυναμίες οι οποίες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Κάτι το οποίο επηρεάζει την ολόκληρη αποτελεσματικότητα αυτών των διαδικασίων εκόλαψης. Όπως επίσης η, η επιλογή των ε, δομών προς επένδυση και χρηματοδότηση δεν έλαβε υπόψη κάποια σημαντικά στοιχεία όπως επίσης ε, όπως ε, οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται, η κατάρτιση του προσωπικού και βεβαίως η οικονομική βιωσιμότητα των επιλεγόμενων δράσεων. Σε μια ειδική έκθεση για τα ταμεία Αλληλεία και για τη στήριξη για τις υδατοκαλλιέργειες καταλήξαμε πως τα έργα τα οποία εξετάσαμε πολλές φορές είχαν επιλεγεί με τον λάθος τρόπο. Για παράδειγμα κάποια έργα είχαν ήδη ολοκληρωθεί όταν είχε ε, ληφθεί η απόφαση ένταξης και σε ένα κράτος ε, είχαμε ε, επιλογή έργων ανάλογα με τη σειρά κατάθεση, το οποίο δεν έλαβε υπόψη ούτε την ποιότητα ούτε ε, και τα άλλα στοιχεία και κάποια τα οποία έφτασαν καθυστερημένα ή εν πάση πτώση μέσα στην προθεσμία αλλά αργότερα αυτά απορρίφθηκαν γιατί δεν υπήρχε πλέον διαθέσιμος προϋπολογισμός και έχουμε και την ειδική έκθεση για τις αεροπορικές υποδομές όπου οι επενδύσεις πολλές φορές δεν ε, ήταν απαραίτητες αποδεικνύονταν μόνο για το 50% των επενδύσεων και γύρω στα 30% από αυτά τα αεροδρόμια δεν ήταν κερδοφόρα και θα είχαν κλείσει εάν δεν υπήρχε συνεχιζόμενη δημόσια στήριξη. Τελικό συμπέρασμα λοιπόν ήταν πως αυτές οι, επιδοτούμενες, ε, οι χρηματοδοτούμενες ευρωπαϊκές ενεργείες δεν, ήταν, δεν πρόσφεραν value for money και για το 2016 στην ειδική έκθεση για τα λιμάνια καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή οι στρατηγικές διάρθρωσης και προώθησης λιμανιών που είχαν υποβάλει τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδιναν τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να έχουμε ε, καλό σχεδιασμό αύξηση δυναμικού με συγχρηματοδοτούμενες δράσεις σε λιμενικές δραστηριότητες και υποδομές που ήταν αναποτελεσματικές και μη βιώσιμες με υψηλό κίνδυνο για 400 εκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν και τα οποία τελικά δεν, δεν ε, χρησιμεύσαν. Πολλές φορές έλειπαν οι διασυνδέσεις με την υπόλοιπη χώρα έτσι ώστε οι λιμενικές αυτές εγκαταστάσεις ουσιαστικά να μένουν αχρησιμοποιητές. Και πολλές φορές η χρηματοδότηση είχε γίνει για το ένα κομμάτι του έργου και αυτή η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τελικά οδήγησε στην επιπλέον ε, δαπάνη εθνικών πόρων σε έργα τα οποία δεν ήταν απαραίτητα. Και αυτά είναι αρκεί για να πρέπει να ξανασκεφτούμε αν αυτά τα έργα θα έπρεπε να έχουν επιλεχθεί και αν πρόσφεραν κάποια προστιθέμενη αξία στους πολίτες. Συστήσαμε να Στιάσουμε στα αποτελέσματα και στις επιπτώσεις το συντομότερο δυνατόν και θα πρέπει στο νομοθέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει το εξή πρώτον στις ε, εταιρικέ σχέσεις να ποσοτικοποιούν τα αποτελέσματα τα οποία θα πετύχει η χρηματοδότηση και να δούμε σε αυτά τα ΣΕΣ εάν υπάρχουν κάποιοι δείκτες κοινών αποτελεσμάτων που να μπορούν να μοιραστούν ανάμεσα στα διάφορα ταμεία για να παρακολουθήσουν την πρόοδο σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν ε, στο πλαίσιο να βασίζεται σε δείκτους απόδοσης που θα λαμβάνει υπόψη αυτά τα, ε, αυτούς τους δείκτες, τους κοινούς δείκτες αποτελεσματικότητας. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν είναι δωρεάν, είναι μεγάλα τα ποσά που χρειάζονται για να συγχρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα και να χρηματοδοτηθούν και κάποια επιπλέον συναφή έργα. Οι εθνικές και οι περιφερειακές κυβερνήσεις και αντιστοίχω τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν αυτή τη δαπάνη που γίνεται από το εθνικό προπολογισμό και να καταλήγουν πως για την απόδοση χρειάζονται δυο για να χορέψουν. Του του τάγκο, όπως λέμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος είναι ο Νίκολας Μάρτης, αναπληρωτής γενικός Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Υποθέσεων Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω στη σημαντική αυτή συνάντηση για ένα τόσο βασικό θέμα. Μου άρεσε πολύ ο τίτλος της συνεδρίας αυτή, επειδή μας κάνει όλους να μας παρακινεί να σκεπτόμαστε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή χρήση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω πως αντικατοπτρίζει αυτό που ήδη κάναμε για το 2014 έως το 2020 με βάση την πρόταση της Επιτροπής η νομοθετική αρχή, δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θέσπισαν για το 2014 έως το 2020 ένα ριζικά διαφορετικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά διαφορετικά και επενδυτικά ταμεία που δημιουργεί μηχανισμούς δημιουργίας επίδοσης βάσει της επιθυμίας να μετακινηθούμε από την απορρόφηση και να προχωρήσουμε σε μια προσέγγιση προσεγγισμένης προσανατολισμένοι στην επίδοση, αλλά πρέπει να ξοδεύονται τα χρήματα για να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Γι' αυτό και δεν αποτελεί εναλλακτική. Και η εμπειρία μας δείχνει πως εάν δεν έχουμε κίνητρα για να δαπανώνται τα χρήματα με εύλογο τρόπο, τότε υπάρχει ο κίνδυνος των καθυστερήσεων. Αυτονόητο είναι επίσης πως είχαμε μεγάλες αυξήσεις των μη χρησιμοποιημένων κονδυλίων που προκάλεσαν μια μόχλευση των εξόδων σε κράτη-μέλη. Γι' αυτό και δεν θεωρούμε πως εδώ προχωρούμε ή απομακρυνόμαστε ή θα πρέπει να απομακρυνόμαστε από κίνητρα, αλλά περισσότερο ότι διασπαλίζουμε την έγκαιρη δαπάνη των χρημάτων και πως έχουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις πως δαπανώνται τα χρήματα με σοφό τρόπο. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης το νέο μηχανισμό αυτό που δεν υπήρχε αλλά δεν αγνοήσαμε το ζήτημα της επίδοσης. Σε καμία περίπτωση είχαμε την αξιολόγηση από τα κρατημέλη και κάναμε μια πολύ ευρεία αξιολόγηση για να δούμε τι απέγινε η χρηματοδότηση αν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια, θα δούμε δύο στοιχεία μακροοικονομικού μοντέλου για να δούμε τι γίνεται με την χρηματοδότηση. Και εκεί βλέπουμε τι απογίνεται η χρηματοδότηση. Το κάθε ευρώ που ξοδεύεται. Αυτό είναι το μοντέλο. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε μια, έναν κατάλογο, δεν θα τον περάσω ένα προς ένα, αλλά έχουμε στοιχεία από την αξιολόγηση για ένα σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, επίσης σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων κτλ. Δηλαδή πήραμε το ζήτημα αυτό στα σοβαρά Κοίταξαμε τι συνέβη και μπορούμε να δούμε επιτεύγματα στον τρόπο δαπάνης της χρηματοδότησης. Αλλά ας κοιτάξουμε το χρονικό διάστημα 14 έως 2020, επειδή η πρόκληση έγκυται ακριβώς εκεί. Αν κοιτάξουμε την επόμενη διαφάνεια, θα δούμε τέσσερα νέα στοιχεία, τα οποία από κοινού συστήνουν το νέο μηχανισμό. Πρόκειται για τον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα που οθεί τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν πως όταν καθορίζουν, όταν λαμβάνουν απο, αποφάσεις για το πώς πρόκειται να χρηματοδοτήσουν κάτι, αυτό να γίνει σε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή, να καθορίζεται το στόχος ο οποίος πρόκειται να επιτευχθεί κατά τη δαπάνη των χρημάτων. για κάθε πρόγραμμα έχουμε ένα πλαίσιο επίδοσης για να έχουμε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της επίδοσης. Χρησιμοποιούμε δείκτες σε ένα χρονοδιάγραμμα και συνέπειες σε περίπτωση μη επιτυχίας των ορόσημων. Σημαντικό είναι να υποθεί πως αυτό γίνεται σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος και όχι σε επίπεδο συμφωνίας. Και πρέπει να γίνει επίσης σε επίπεδο επιχειρησιακού προγράμματος, επειδή σε αυτό το επίπεδο λαμβάνονται οι αποφάσεις και σε αυτό το επίπεδο μπορούν να οριστούν οι συγκεκριμένοι στόχοι που χρειάζονται για να μπορέσουν να καθοριστούν ρεαλιστικοί δείκτες για αυτά. Επίσης έχουμε έναν πιο έντον, μια πιο έντονη υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να παρέσχουν αποδεικτικά στοιχεία πως έλαβαν τις κατάλληλες αποφάσεις εξ αρχής και έχουμε και αρκετές προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν πως υπάρχουν τα προαπαιτούμενα για να διασφαλιστεί η δαπάνη των χρημάτων στο κατάλληλο πλαίσιο. Έτσι έχουμε αφενός κανονισμούς, οδηγίες, αλλά ακόμα πιο σημαντικό χρειαζόμαστε τις κατάλληλες στρατηγικές. Αν θέλουμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, μια έξυπνη στρατηγική εκπαίδευση κτλ οι αποφάσεις για την επιλογή επιχειρήσεων δεν πρέπει να γίνονται με τυχαίο τρόπο, αλλά σε συνδυασμό με μια στρατηγική η οποία θα δείχνει πως η διαδικασία επιλογής είναι η κατάλληλη. Στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα, θα δούμε τον κύριο πυρήνα του ζητήματος. Έχουμε ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων όταν κατά τη φάση προγραμματισμού σχεδιασμού. Όταν η αφετηρία είναι η προσπάθεια επίτευξης στόχων. Τα κράτη-μέλη δηλαδή πρέπει να ορίσουν τους εκάστοτε στόχους, να ταυτοποιήσουν τους δείκτες και στη συνέχεια να επανέλθουν στις επιχειρήσεις που θα χρηματοδοθούν. Και στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε έναν απλό τρόπο να το εξηγήσουμε. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διερωτηθούν σχετικά με τρία ζητήματα. Τι πρέπει να αλλάξει μέσω της επένδυσης, πώς θα μετρηθεί αυτή η αλλαγή και ποιες δράσεις μπορούν να συνεισφέρουν στην αλλαγή την οποία επιθυμώ. Υπάρχει ένας απλός τρόπος για να γίνει όλο, όλος, όλη αυτή η προσέγγιση κάτι απτό. και το πλαίσιο της επίδοσης. Έχουμε τον τρόπο ίχνηλάτησης εδώ μέσω βασικών δικτών, οι οποίοι συνδέονται από τη μία με κίνητρα και αφετέρου με δυνητικές κυρώσεις απώλειας της χρηματοδότησης σε περίπτωση που οι στόχοι δεν επιτευχθούν στο τέλος του προγράμματος. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως ξεχνούμε τις τυπικότητες οι οποίες θα, θα συνεχίσουν να είναι σημαντικές και χρειάζονται για τον έλεγχο των δαπανών κατά την ε, διάρκεια της περίοδου και είμαι σίγουρος πως θα έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Συμπεραίνοντας λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα στο οποίο ένα κράτος μέλος μπορεί ακόμα να απολέσει τη χρηματοδότηση λόγω μη χρήση τη και πιστεύουμε πως ο μηχανισμός αυτός είναι δικαιολογημένος για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη δαπάνη. Έχουμε όμως επίσης μηχανισμούς κινήτρων που σχετίζονται με την επίδοση. Τα κράτη μέλη επιτυχάνουν δηλαδή τα ορόσημα που καθορίζονται και έχουμε και τα εργαλεία της αναστολής τόσο για την μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων όσο και για την μη επίτευξη των οροσίμων. Επιτύχαμε πιστεύω με την βοήθεια και στεναρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα νέο πλαίσιο το οποίο αποτελεί μια μεγάλη πρόοδο και το βλέπουμε ήδη στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σε έναν παλιό γνώριμο, τουλάχιστον ε, όσον αφορά το όνομα, στον κύριο Βαν Ρομπέι, ο οποίος έρχεται από το Βελγικό ε, Επιμελητήριο Τώρα πρέπει να σας πω, εμείς δεν τα έχουμε καταλάβει καλά. Ε, ποιο επιμελητήριο κάνει τι. Για τη Βαλονία, με τη Βαλονία ασχοληθήκαμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Ε, ίσως λοιπόν πρέπει να εξηγηθούν ορισμένα πράγματα. Σας καλωσορίζουμε θερμά. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Δυστυχώς ε, δεν χρησιμοποιεί μικρόφωνο ο μιλητής. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ είμαι πρόεδρος ε, του Βελγικού Προεδρικού Επιμελητηρίου. Ομιλώ ε, εξ ονόματος του Βελγικού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Οικονομικών ε, Υποθέσεων και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχει κανείς ε, κατά νου, να ξέρει κάτω ποιο πρίσμα κρίνεται η Ευρώπη. Εμείς καταθέσαμε τον προϋπολογισμό μας και περιμένουμε την κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κατά πόσον δηλαδή σεβόμαστε, τηρούμε το 3%, μήπως χρειάζεται να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το 2018. Βάση περιπτώσει, ε, θέλουμε να μετριάσουμε λίγο τις ε, φιλοδοξίες μας, αν δεν επιθυμούμε να καταλήξουμε σε διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος. Οι προϋπολογισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τους ε, προϋπολογισμούς ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, είναι σημαντικό την ε, ε, δημοσιονομική μας πολιτική να την εξετάζουμε κάτω από το ίδιο πρίσμα. Ε, γιατί τελικά όλοι έχουμε δεσμευτεί να καταθέτουμε και να έχουμε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Έχουμε δεχτεί το 3%. Μέσω πρόθεσμα λοιπόν Θέλω να ελπίζω ότι θα κατορθώσουμε να καταργήσουμε πλήρως τα ελλείμματα για να μην αυξηθεί περαιτέρω το χρέος μας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό στο μέλλον σε συναντήσεις ε, όπως αυτή που λαμβάνει η χώρα σήμερα, σε τέτοιου είδους συναντήσεις, να τονιστεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια οφείλουν να ελέγχουν αυστηρότερα την ε, ελεγκτική εξουσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό της προπολογισμό, τα δικά της κονδύλια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Επιτροπές Προϋπολογισμού οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγχουν τους προϋπολογισμούς για το τι πραγματικά υλοποιείται και έναν προϋπολογισμό μπορεί κανείς να τον κρίνει μόνο εφόσον ελέγχει αυστηρά την εφαρμογή αυτού του προϋπολογισμού. Το 2018 ε, θα χαρακτηρίζεται πάλι από οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ως εκ τούτου είναι απολύτως απαραίτητο ε, να ελέγχονται τα κονδύλια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε τελική ανάλυση είναι χρήματα φορολογουμένων και ο φορολογούμενος πρέπει να γνωρίζει πώς γίνεται η χρήση των κονδυλίων του. Μηδενική ανοχή, αυτό είναι σημαντικό. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο, ένας ε, ευρωπαϊκός θεσμός ε, ελέγχου και οι διοικητικές υπηρεσίες του ελεγκτικού συνεδρίου καταβάλουν προσπάθειες να εντοπίζουν το ποσοστό σφάλματος. Δηλαδή πόσα κονδύλια χάνονται, ίσως γιατί δεν γίνεται σωστή εφαρμογή του προϋπολογισμού. Ε, νομίζω βελτιώσεις μπορεί κανείς να επιτύχει αν ε, αντιμετωπιστούν σωστά τα υψηλά ποσοστά σφάλματος, κυρίως σε συγκεκριμένες χώρες. Η ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου εξακολουθεί να δείχνει ότι το ποσοστό σφάλματος υπερβαίνει το 5%. Πριν από κάποια χρόνια μιλάγαμε για 10%. Άρα δηλαδή διαπιστώνουμε πλέον μια ουσιαστική βελτίωση. Παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να υπάρξουν βελτιώσεις, να καταπολεμηθούν οι απάτες, να επιδιώξουμε βελτιώσεις γενικότερα. Και αν θέλετε, τα στοιχεία του προπολογισμού ε, να βρίσκονται πιο κοντά στην πραγματικότητα. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι μέσω πρόθεσμα η διαχείριση του προπολογισμού και η έλεγχη από τα κράτη-μέλη είναι κάτι το σημαντικό. Μία κακό κείμενη πολιτική πρέπει να διορθώνεται τη στιγμή μάλιστα που μπορεί να αποτελεί φυτόριο για αντιευρωπαϊκά αισθήματα. Αν λοιπόν έχει κανείς την αίσθηση ότι προκύπτει κακή διαχείριση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καταλήγει ίσως κανείς και στο συμπέρασμα ότι γενικά η Ευρώπη δεν λειτουργεί σωστά, ότι δεν είναι σωστή η έλεγχη. Με λίγα λόγια οφείλουμε να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να αντιδράσει και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την αξιόπιστη πολιτική που μας ε, κατατέθηκε. Το 2016 θα λάβει τελική μορφή η διαμόρφωση των διαρθρωτικών ταμείων και θα καταβάλουμε προσπάθειες να ελέγξουμε την κατάσταση. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαλλάσσονται, αλλά νομίζω ότι ξεκολουθεί να υπάρχει πετιότητα που ανάγεται στην Επιτροπή Σαντέρ για το ότι τα, ε, το κοινοβούλιο ξεκολουθεί να συμπεριφέρεται ως συμπεριφέρεται. Τα εθνικά κοινοβούλια θεωρούν ότι θα πρέπει και αυτά και τα περιφερειακά κοινοβούλια να συμμετέχουν στους ελέγχους. Όμως ε, εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχει ψηλό ποσοστό σφάλματος, εκτεταμένες απάτες, εφόσον διαπιστώνεται όλα αυτά, τίθεται αυτόματα και το ερώτημα μήπως ε, θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική για την επιδίωξη βελτιώσεων. Δηλαδή τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στοχευμένα. Αυτό το use it or lose it αν δεν χρησιμοποιήσει δηλαδή, τα κονδύλια θα χαθούν. Αυτό πρέπει πια να σταματήσει. Η δημοσιονομική πολιτική είναι καθοριστική σημασία για την ε, αξιοπιστία, εμπιστοσύνη από πλευράς πολιτών. Ε, στόχος μας λοιπόν θα πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη βελτίωση. Διάφορα κράτη-μέλη ε, έχουν αποκεντρωμένες αρμοδιότητες για τη διαχείριση των κονδυλίων, όμως η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων μπορεί να είναι και αρνητική. Αν τελικά οι αρμοδιότητες δεν έχουν καθοριστεί και δεν έχουν επιμεριστεί σωστά στα τρία επίπεδα, τότε γίνεται και κακή διαχείριση κονδυλίων μία συνεδρίαση η οποία όπως αυτή σήμερα λαμβάνει σήμερα χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μια τέτοια συνεδρίαση καταδεικνύει ότι μπορούμε να εργαζόμεθα αποτελεσματικά σε διάφορα επίπεδα και ειδικά όσον αφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό, νομίζω ότι ε, οι ευθύνε είναι σαφείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, μάλλον να το πω το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζουν μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κατά πόσον ο προϋπολογισμός είναι ικανοποιητικό και τα δύο αυτά όργανα εκ των υστέρων καλούνται να ελέγξουν. Άρα δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε είναι και έλεγχος και πολιτικό όραμα εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σε σχέση με το μέλλον. Καταρχήν, ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή προϋπολογισμός και επταετή δημοσιονομικά προγράμματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια προοπτική, από την άλλη όμως να μην είμαστε άκαμπτοι, να μην εγκλωβιζόμαστε σε αγκυλώσεις, να υπάρχει μια ευελιξία, όπου βέβαια ε, για όλα αυτά χρειαζόμαστε ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε κατευθυνόμενη οικονομία της αγοράς με βάση το σοβιετικό μοντέλο, όχι μακροπρόθεσμο όραμα με ε, αυθόρμητες και ε, παρεμβάσεις. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ε, συμφωνούμε πολύ ε, με αρκετά από αυτά που είπατε, θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Από την Πολωνία. Χαίρομαι που ήρθατε κύριε Πόλνιτς. Ε, δεν περίμενα ότι θα έρθατε. Ήξερα μόνο ότι δεν θα έρθει κάποιος αδελφός σας. Σας καλωσορίζουμε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, Εκπροσωπώ εδώ την, ε, το Πολωνικό Κοινοβούλιο και μάλιστα εκπροσωπώ την Ανατολική Πολωνία, όπου είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες χάρη στα όσα προέσφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα όμως πάρα πολλά πρέπει να γίνουν και εδώ χρειάζεται να τονίσω πως εμείς είμαστε υπέρ μιας πιο αποτελεσματικής χρήσης των κονδυλίων που φτάνουν στην περιοχή μου από τις Βρυξέλλες. Παράλληλα όμως είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε πως η κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που να είναι πιο ε, ευνόητος από τον Ευρωπαίο πολίτη. αυτό που είπαμε για τα γεωργικά ταμεία. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές πως η νέα πρόκληση δεν είναι μόνο ότι τα χρήματα χρειάζονται για τοπικούς, να καλύψουν τους τοπικούς στόχους, αλλά για να έχουμε χαμηλότερες εκπομπές, για καλύτερη παιδεία, για μια καινοτόμο οικονομία και για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιθυμώ επίσης να πω πως οι μεταρρυθμίσεις είναι βεβαίως απαραίτητες, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί προσεκτική τη στιγμή που τις ε, εισάγουμε γιατί ε, δεν θα πρέπει η νέα μεταρρύθμιση να οδηγήσει στην απώλεια ε, παλαιών εκτιμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να ευθυγραμμιστούμε με τα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με την κατάλληλη και την αποτελεσματική χρηματοδότηση αυτών των έργων. Ευχαριστώ πολύ για όσα είπατε. Αν κάποιος θέλει το λόγο, τότε χρειάζομαι ένα, μια μπλε σελίδα Ανάλογα με τα ταμεία διαφέρει η κατάσταση. Για το Αγροτικό Ταμείο μιλήσαμε πριν. Έχουμε την Όσον αφορά τι διοικητικέ αρχέ στο, στο Γεωργικό Ταμείο, έχουμε μια παρόμοια κατάσταση, αλλά και πρόσθετα προβλήματα λόγω τη φύση των διαφορετικών ταμείων. Και η φύση είναι πως υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα στο σύστημα αυτό, ίσως υπερβολικά χρήματα. Μόνο έτσι είναι δυνατόν η συσσόρευση τεράστιων ποσών τα οποία δεν εφαρμόζονται, δεν, ξοδεύονται σε, μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων. Όταν επενδύουμε εμείς χρήματα θεωρούμε δεδομένο πως πρέπει να δαπανώνται τα χρήματα αυτά. Αλλά έχουμε ένα υπόλοιπο στον προπολογισμό το οποίο μεταβιβάζεται από χρονιά σε χρονιά και πλέον χρειαζόμαστε πάρα πολύ για να κλείσουμε ε, οριστικά ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να διαρκέσει έως και 20 χρόνια. Αυτό μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο. Και στο τέλος της περίοδου, όταν καταπίπτουν τα χρήματα, τότε αρχίζουν τα προβλήματα καθέφτα. Βλέπουμε πως πολλά κράτη-μέλη ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη χρήση των χρημάτων με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς να ελέγξουν εάν το πρόγραμμα το εκάστοτε πρόγραμμα χρειάζεται μπορούμε να μιλούμε όλο το βράδυ. Μπορώ να διηγηθώ ιστορίες για προγράμματα τα οποία δεν χρειαζόταν κανείς. Γι' αυτό και από πλευρά μα θα ήταν αναγκαίο τα ευρωπαϊκά χρήματα αυτά να τοποθετούνται πιο στοχευμένα και καλύτερα για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πιστεύω πως χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες προϋποθέσεις από ό,τι το κάνουμε σήμερα. Πιστεύω πως αυτή είναι η τάση την οποία διαβλέπουμε. Επειδή τα χρήματα αυτά αποκτούν όλο και περισσότερη αξία, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν όλο και λιγότερα. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας παροτρύνω, επειδή το ερώτημα τι αποτέλεσμα έχει Πού είναι η προστιθέμενη αξία, τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Το ερώτημα αυτό είναι σημαντικό για εμάς και θα μας απασχολήσει επίσης κατά το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο στη συζήτηση. Με αντίστροφη σειρά θα ήθελα να ζήσω από τον κύριο Μάρτι να μας πει κάποια πράγματα για τις ερχόμενες δημοσιονομικές περιόδους. Ο κύριος Λαζάρου θα μας μιλήσει λίγο σύντομα για τα διαφορετικά ταμεία και το λόγο θα λάβουν επίσης τα εθνικά κοινοβούλια και θα ήθελα κυρία Βαλουρόμπου να σας ζητήσω επειδή βλέπουμε συχνά πως στα κράτη-μέλη υπάρχουν συνταγματικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την απορρόφηση της χρηματοδότησης. Στην περίπτωση της Ισπανίας μπορούμε να γράψουμε ένα ολόκληρο βιβλίο σχετικά με αυτό που προέρχεται από την ομοσπονδιακή φύση του κράτους. Και η Γερμανία είναι ομοσπονδιακό κράτος αλλά αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα. Γι' αυτό και θα ήταν ωραίο να ακούγαμε από την οπτική σας γωνία κάτι από την οπτική γωνία του Βελγίου. Η περιφέρεια, η περιφέρεια των Βρυξελών Αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αρχέ του έτου είχαν λυθεί τα προβλήματα αυτά. Ελπίζουμε η κατάσταση να παραμείνει ω έχει ω το τέλο του χρόνου. Ποιε δυνατότητε υπάρχουν από τη δική σα σκοπιά να επέμβει κανεί σε εθνικό επίπεδο, κύριε Μάρτιν. Σας ευχαριστώ και πάλι κυρία Πρόεδρε ίσως ε, κάποια σημεία στα οποία θα έπρεπε να επανέλθω και τα οποία ακούστηκαν και στη σημερινή συζήτηση. Καταρχήν τα ποσοστά σφάλματος που προέκυψαν ως θέμα δεν με εκπλήσουν. Πολύ συχνά συζητάμε για το ποιο είναι το ποσοστό σφάλματος στην Επιτροπή σας στα πλαίσια της ε, πολιτικής συνοχής και διαρθωτικών ταμείων και μάλιστα κάποιο είπε πως το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεση για την περίοδο του 2013 διαπίστωσε πως το ποσοστό σφάλματος που καθόρισε είναι γύρω στο 5 με 6%. Θα ήθελα λοιπόν Να δώσω το γενικότερο πλαίσιο με στο οποίο αυτό προέκυψε και αυτό βρίσκεται και στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και στην ετήσια έκθεση την οποία ε, προετοίμασε η δική μας Γενική Γραμματεία, η Γενική Διεύθυνση. Να σας πω πως όταν φτάσουμε στο τέλος της αλυσίδας ελέγχου το ποσοστό αυτό αλλάζει. Οπότε αυτό το οποία εμείς ε, βρίσκουμε βασιζόμενοι στις ελεγκτικές δραστηριότητες των εθνικών αρχών είναι ένα επικυρωμένο ποσοστό σφάλματος γύρω στο 3% και μετά πρέπει να λάβει κανείς υπόψη τις διορθωτικές ε, δράσεις που αναλαμβάνονται και όπως σας είπα η μεθοδολογία που μας οδηγεί στον καθορισμό αυτό μας βοηθά στο να καταλήξουμε σε μια ε, αξιοπιστία πως το υπολοιπόμενο ποσοστό σφάλματος είναι κάτω από το 2%. Αυτό βέβαια ξεκαθαρίζει περισσότερο κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της περίοδου 2013 και όταν κλείσουν όλα πια και καταλήξουμε στο τελικό νούμερο θα σας ενημερώσουμε. Το άλλο πολύ σημαντικό στο οποίο αναφέρθηκα εδώ εντάχει είναι πως κάναμε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσουμε αυτή την αξιοπιστία για το θέμα της συμμόρφωσης, για την πολιτική συνοχής, για την περίοδο 14-20. Αυτό θα μας βοηθήσει να είναι μεγαλύτερη η αξιοπιστία για το ποιο είναι το υπολοιπόμενο ε, ποσοστό σφάλματος, γιατί θα εξετάζουμε μια δωδεκάμενη περίοδο απομονωμένα από τις υπόλοιπες και θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το ποιο ήταν το ποσοστό σφάλματος που απομένει εκεί και μέσω αυτού του συστήματος πιστεύουμε πώς θα μπορούμε να αποδεικνύουμε πως αυτό το άλμα που κάναμε από το 2000-2006 στην περίοδο 7-13 που μειώσαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό το ποσοστό σφάλματος θα πάει ένα βήμα παρακάτω και θα έχουμε όντως αυτή την αξιοπιστία που θα προσφέρει την εμπιστοσύνη ε, στο κοινό που θα ξέρει πως τα ταμεία αυτά ελέγχονται. Τώρα, κάποιος με ρώτησε τι γίνεται με το διοικητικό δυναμικό ε, για να μπορούμε λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί στα όσα παραδίδουν αυτά τα ταμεία, χρειάζεται να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να ενισχύσουμε τη δική τους, ε, το δικό τους δυναμικό. Και αυτό γίνεται και μέσω αιρεσιμότητα που αποτελεί τον τρόπο για την οικοδόμηση δυναμικού αλλά και μέσω τη τεχνική βοήθεια και της συναφών δράσεων ε, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη στήριξη άλλων θεσμών. Όλα αυτά είναι στοχευμένα για τα κράτη-μέλη που έχουν λιγότερο ή μάλλον πιο αδύναμε δικήσει και που χρειάζονται αυτή την επιπλέον στήριξη έτσι ώστε να στήσουν για παράδειγμα αυτή τη στρατηγική για την ευφύ εξειδίκευση, Smart για παράδειγμα. Και νομίζω ότι υπάρχει ευρύτατη στήριξη με κάποιες πειραματικές δράσεις σε κάποιες περιοχές έτσι ώστε να είναι πολύ πιο απτές οι προσπάθειες που κάνουμε, να είμαστε πιο κοντά στις εθνικές περιφερειακές διοικήσεις για να προχωρήσουμε κάπως προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, για τις απεντάξεις. Όταν μιλήσουμε για το τι έγινε για την περίοδο 7-13, θα δείτε πως για το ΕΤΠΑ και για το Ταμείο Συνεχής και για την απένταξη, δηλαδή τα ποσά τα οποία χάθηκαν για πάντα, μιλάμε για το ένα περίπου δις ε, από τα 270 δις που ήταν το συνολικό ποσό. Άρα λοιπόν, εντάξει, τους τελικούς λογαριασμούς θα τους κάνουμε όταν κλείσουν τα προγράμματα, αλλά η τελική ημερομηνία για την κατάθεση των ε, ε, εγγράφων κλεισίματος είναι ο Μάρτιος του 2017 και αυτή τη στιγμή μόνο δύο-τρία κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον υποκίνδυνο να χάσουν ένα υψηλό ποσό. Άρα λοιπόν ο μηχανισμός απεντάξεων έχει αυξήσει την απορροφητικότητα και την απορρόφηση, με συγχωρείτε, και είναι ένας καθόλου νόμιμος τρόπο να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, εξασφαλίζοντα παράλληλα τον σεβασμό των κανόνων και την απόλυτη συμμόρφωση έτσι ώστε να επινηχάνουμε και τα κατάλληλα αποτελέσματα. Τώρα, τι οδηγεί την απόδοση ε, στο επόμενο στάδιο, η διαφάνεια. Και δεν χρειάζεται μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει και να επιπτεύει ότι γίνεται καλή χρήση των κονδυλίων. Θα πρέπει αυτό να είναι δυνατόν και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. και νομίζω ότι σε αυτό θα μας βοηθήσουν και οι Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι πολίτες. Εν ώψη του 2020 λοιπόν θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και αυτό ε, μπορεί να γίνει μέσω των πλατφόρμων ανοιχτών δεδομένων όπου οποιοδήποτε μπορεί να πάει ε, online και να δει τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τι έχει υπογραφεί ποιε είναι οι προθέσει για τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν και μετά να παρακολουθεί την χρήση των κονδυλίων έτσι ώστε να γνωρίζουμε από τα κονδύλια αυτά τι αποκομίζουμε. Τα κράτη-μέλη λοιπόν μέσω των ετησίων εκθέσεων που υποβάλλουν δίνουν αυτά τα δεδομένα τα οποία μετά είναι απολύτως προσβάσιμα έτσι ώστε να είναι ορατά και να μπορούν να τα εξετάσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένας από τους παράγοντες που θα μας βοηθήσουν στο να εστιάσουμε στην απόδοση με τη χρηματοδότηση. Τώρα, ας ατενίσουμε λίγο το μέλλον. Βρισκόμαστε ακόμα σε μια πρώιμη ε, φάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μετά το 2020 εποχή και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως προκύπτει από τις συζητήσεις που κάναμε για τον προϋπολογισμό που θα εστιάζει στις, ε, στους στόχους και από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανδιάμεση Αναθεώρηση πως ο στόχος μας θα είναι να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτά που έχουν επιτευχθεί το 14-20 και να χρησιμοποιήσουμε τα τεκμήρια που θα έχουμε από αυτή τη γενιά έργων για να εντοπίσουμε τι λειτουργήσε και τι χρειάζεται να ενισχυθεί παραπάνω. Και κυρίως για την πολιτική συνοχή, να σας πω πως αυτά τα πλαίσια η αιρεσιμότητα μοιάζει να είναι ένα εργαλείο το οποίο παραδίδει χρήσιμα αποτελέσματα και να δούμε πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε και να εξελίξουμε περαιτέρω αυτή τη δυνατότητα. Βεβαίως κρίσιμο είναι κρίσιμο είναι να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η απλούστευση λοιπόν, και πολλοί θεωρούν πως τα κράτη-μέλη ε, δεν μπορούν να κάνουν αυτή την αποκοινού διαχείριση με τον κατάλληλο τρόπο, το shared funding δηλαδή. Οπότε για την ενδιάμεση αναχυθεώση να σας πω πως τα συμπεράσματα ε, είναι πως όπου μπορούμε πρέπει να προχωρήσουμε με το τρέχον πλαίσιο, αλλά παράλληλα πως θα χρειαστεί και ένα άλμα που θα μας οδηγήσει πολύ πιο μακριά η ευελιξία αναφέρθηκε και αυτό είναι θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τις σκέψεις για τη μετά το 2020 εποχή, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο σύνδεσμος με την οικονομική διακυβέρνηση με τρόπο που θα απηχεί τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Αυτά λοιπόν. Αυτοί είναι οι συλλογισμοί των επόμενων μηνών που θα οδηγήσουν σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τα τέλη της επόμενης χρονιάς. Και για την πολιτική συνοχή να σας πω ότι θα έχουμε και κάποιους ακρογωνιαίους λίχους, κάποια ορόσημα σε όλη τη διαδικασία. Έχουμε το φόρουμ για τη συνοχή του χρόνου τον Ιούνιο, που θα είναι μια ευκαιρία για να γίνει μια διαβούλευση και μια συζήτηση για κάποια από τα κομβικά ζητήματα, όπως επίσης και η έκθεση για τη συνοχή που θα δημοσιευθεί το δεύτερο εξάμεινο της επόμενης χρονιάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω η συζητήση ήθελε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ακριβώς ε, επειδή έχουμε κοντά μας τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Περιφερειών, κανένας εξ αυτών δεν αμέλησε να πει το πόσο σημαντικά είναι τα διαρθρωτικά ταμεία για τις ε, περιφέρειες και για τα κράτη-μέλη. Τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων. Όλοι το είπαν αυτό. Όμως αυτό που ανησυχεί λιγάκι είναι το πώς χειρίζονται τα κράτη-μέλη αυτά τα κονδύλια. Δηλαδή, ήδη τρέχει περίοδος του 2014. Όμως ε, τέλος του 2015 βλέπουμε ότι υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών ήδη από την προηγούμενη περίοδο για το 2013 πάνω από 23 δις και αυτά είναι κονδύλια τα οποία έχουν υπολογιστεί με βάση την στήριξη προγραμμάτων της προηγούμενης περίοδου. Όλα αυτά λοιπόν ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρόκειται για χρήματα τα οποία τα έχουν δαπανίσει τα κρατημέλη και κανονικά πρέπει αυτά τα χρήματα να λείπουν από τους προϋπολογισμούς τους. Παράλληλα όμως διαπιστώνουμε μια τεράστια καθυστέρηση κατά την έναρξη της νέας περίοδου. Διαπιστώνουμε ότι το 1 πέμπτο των κρατών μελών έχουν ορίσει τους οργανισμούς πληρωμής για την εκαθάριση. Υπήρξε μια τεράστια καθυστέρηση στον ε, καθορισμό των ε, φορέων για συνεργασία και αυτό ήταν προϋπόθεση για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Τώρα αυτό επιβεβαιώθηκε κατά 100%. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει η εργασία για συγκεκριμένα προγράμματα, όμως ήδη έχουν περάσει τρία χρόνια της τρέχουσας περίοδου. Και ο κύριος ε, Μάρτιν είπε ότι το 18-19 ήδη για τότε θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης και καθάρισης, γιατί με βάση τα αποτελέσματα τότε ε, με βάση αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και το απόθεμα το οποίο έχει κρατηθεί. Σας τα λέω αυτά για να σας δείξω ότι εδώ ελοχεύουν πάρα πολλοί κινδύνοι. Μα αν είναι όλα τόσο σημαντικά θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο σοβαρή εργασία, να εφαρμόζονται τα προγράμματα, ε, γιατί αν δεν γίνεται αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι Υπάρχουν τόσες πολλές απαιτήσει από τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό που τελικά δημιουργούνται και πάρα πολλοί περιορισμοί. 80% των κοντιλίων μεταφέρονται με τη μορφή διαρθρωτικών κοντιλίων στα κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου λοιπόν, ίσως θα πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσο μπορούμε να συνεχίσουμε την πολιτική συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική με τη μέχρι τώρα μορφή της και κατά πόσο είμαστε σε θέση να τη συνεχίσουμε με την μέχρι του μορφή της. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα σε εκείνους που είναι οι δικαιούχοι, οι αποδέκτες, εκεί δηλαδή που εφαρμόζουν τα προγράμματα και ό,τι γίνεται εκεί είναι δική τους ευθύνη, ανάμεσα σε αυτούς και στους άλλους που έχουν συγκεκριμένους ε, στόχους, ε, δηλαδή το ευρωπαϊκό επίπεδο συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, αν υπάρχουν ε, εμπόδια για να εφαρμόζονται όλα αυτά όπως πρέπει, νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όχι τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια να αντιμετωπίσουμε και πάλι το ίδιο πρόβλημα, μόνο που το ίδιο πρόβλημα θα έχει διωγκωθεί για τον προπολογισμό του 2017 που είναι στραπατσαρισμένος λόγω των ε, εξελίξεων που έχουν προκύψει έχουν μειωθεί κατά πολύ τα διαρθρωτικά κονδύλια Ξέρετε γιατί, γιατί περιμένουμε ότι δεν θα υπάρχει σχεδόν καθόλου εκαθάριση προγραμμάτων από την τρέχουσα περίοδο. Υπάρχουν ήδη κάποιες καθυστερήσεις, αυτά όλα μετατίθενται στο μέλλον και πρέπει να συζητήσουμε από αυτού κατά πόσο μπορούμε από κοινού, θέλουμε ή μπορούμε ακόμα να αναχαιτήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Μπαν με μετά στον κύριο Λαζάρου και μετά θα πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακό κράτος με πολλές αρμοδιότητες για τα ομοσπονδα κρατήδια της Βαλονίας, της Φλάνδρας και των Βρυξελών. Και στην περίπτωση της ΣΕΤΑ είδαμε πως αυτό το Σύμφωνο Ελεύθερου Εμπορίου έγινε αποδεκτό από τις τρεις περιφέρειες, και, αλλά όχι από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Δηλαδή υπάρχει ανεξαρτησία των περιφερειών. Στη Γερμανία έχουμε το υποχρεωτικό Ομοσπονδιακό Δίκαιο, κρατηδιακό δίκαιο, Εάν καταλαβαίνω καλά, υπερισχύει το ομοσπονδιακό δίκαιο του περιφερειακού, το οποίο στο Βέλγιο δεν είναι έτσι οι περιφέρειες εκεί έχουν κυρίαρχα δικαιώματα, το οποίο ισχύει και για τα διαφορετικά ταμεία, τα οποία αποφασίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, όπου και γίνεται και η διαχείρισή τους η φλαμανδική οικονομία αποφασίζει για ζητήματα οικονομίας και θέσεων εργασίας και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Η, η ομοσπονδιακή, δηλαδή η εθνική κυβέρνηση, έχει λίγα να πει σε σύγκριση με τις περιφέρειες στο Βέλγιο οι συνιστώσεις περιφέρειες διαφέρουν πέρα αυτού κατά πολλού. Στη Βαλονία η διαφορετική ανεργία είναι πολύ ψηλή. Έχουμε μια περιφέρεια σε μια καθοδική πορεία που αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να προσελκύσει τεχνολογικές επιχειρήσεις, να ασκήσει μια επιχειρηματική και κοινωνική πολιτική στη Βαλονία σε σύγκριση με το υπόλοιπο Βέλγιο ε, έχουμε μια πολύ αδύναμη δομή. Πρόκειται για την οικονομικά πιο αδύναμη περιφέρεια του Βελγίου με την υψηλότερη ανεργία και τα υψηλότερα διαφορετικά προβλήματα. Στη Φιλάνδρα η κατάσταση είναι διαφορετική. Εκεί η γεωργία είναι πολύ σημαντική αποτελεί επίσης περιφερειακή, δηλαδή κρατηδιακή αρμοδιότητα, η οποία είναι αρκετά μεγάλη και αναλογεί στα επιμέρους κρατήδια, στις περιφέρειες. Εκεί αποφασίζουν επίσης οι περιφερειακές κυβερνήσεις, ενώ το Εθνικό, το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο δεν έχει την αρμοδιότητα να εκφέρει κάτι περισσότερο από μία άποψη. Επειδή στην, στο Βέλγιο η ανεξαρτησία των περιφερειών είναι πολύ έντονη και αφορά επίσης τη χρηματοδότηση των, από τα διαφορετικά ταμεία που αποφασίζεται στα περιφερειακά κοινοβούλια του Βελγίου. Γι' αυτό και υπάρχουν όλο ένα και πάλι συζητήσεις για την αποτελεσματικότητα για την χρήση το, της χρηματοδότησης των διαθαρτικών ταμείων πολλές φορές δεν γίνεται με αποδοτικό τρόπο ή με τρόπο που να έχει νόημα, αλλά τα τελευταία έτη τουλάχιστον γίναμε πιο επιλεκτικοί. εστιάζοντας περισσότερο, μέσω κριτηρίων τα οποία εστιάζουν περισσότερο στην επίδοση. Αλλά όπως είπα, το Εθνικό Βελγικό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα κρίση τη αποτελεσματικότητα, τη αποδοτικότητα τη χρηματοδότηση των διαθροτικών ταμείων, η οποία αρμοδιότητα βρίσκεται στις περιφέρειες, οι οποίες είναι κρατήδια του Βελγίου, συνιστώντα κρατήδια του του Βελγίου, τα οποία όμως έχουν αρμοδιότητες οι οποίες υπερβαίνουν την εθνική κυβέρνηση. Υπάρχουν έντονες τάσεις ανεξαρτητοποίησης, υπάρχουν μάλιστα και αποσχιστές, αλλά Εάν κοιτάξει κανείς τις δημοσιονομικές εξουσίες, τότε αυτές των κρατηδίων, δηλαδή των περιφερειών, είναι σχεδόν οι διπλάσιες από αυτές της Ομοσπονδιακής Βελγικής Κυβέρνησης. Εάν κοιτάξει εάν δεν λάβει κανείς υπόψη το χρέος των περιφερειών. Αυτό ισχύει επίσης για τη χρήση της χρηματοδότησης των κονδυλίων. Ελπίζω να απάντησα σωστά την ερώτησή σας. Um, Πολύ ωραία αυτά που μας είπατε θα τα λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, στο θέμα της αύξησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Και δεν θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαζάρου για να μας κάνει παρατηρήσεις για αυτό το θέμα και να μας εισαγάγει ε, στο επόμενο θέμα που είναι ένα νέο μοντέλο ε, συνεργασίας ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα θέμα το οποίο είναι το εξής. Από τώρα και στο μέλλον ε, θα πρέπει να υπάρχει μία επιτάχυνση διότι διαπιστώνονται καθυστερήσεις και νομίζω ότι και τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουν το θέμα. Εμείς, επί του θέματος, θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες για να φτάσουμε πιο κοντά στην ε, μία και μόνο, στην ενιαία προσέγγιση τα, οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών ε, θα πρέπει να έχουν εξετάσει, να έχουν ελέγξει τις αιτήσεις ακαθαρίσεις πριν εμείς ε, περάσουμε στο δικό μας τον έλεγχο και ε, θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί συλλογικά μέτρα. Νομίζω με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε μόνοι μας να περιορίσουμε το θέμα της ε, δουλειά που να κάνουμε για να διαπιστώσουμε τη συμμόρφωση. Κάτι άλλο, τα χρηματοψηφιακά εργαλεία. Για να αποφύγουμε το να μην ε, εκταμιεύονται κονδύλια στους αποδέκτες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα χρήματα τα οποία δαπανώνται θα πρέπει να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδείξεις ότι τα κονδύλια αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και στην υποδομή. Μέχρι τώρα ε, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Υπολείπονται λοιπόν ακόμα πάρα πολλά επί του θέματος. Πάμε τώρα σε ένα νέο μοντέλο. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές για να επιτύχουμε καλύτερα την ενιαία προσέγγιση. Του χρόνου θα πρέπει να δούμε κατά πόσον η Κομισιόν μπορεί να ε, επωφεληθεί από, τους, από τις δαπάνες. Επίσης, να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά τη συμμόρφωση. Ε, εμείς θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το όλο θέμα στην, ε, της έκθεσή μας θεωρούμε ότι τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να συμβάλλουν διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες δεν θα είναι ε, περίπλοκοι, ε, να στηρίζονται τα αποτελέσματα ε, και να υπάρχει αξιοπιστία. Πώς μπορούν να επιτευχθούν όλα αυτά. Ε, όπως σας είπα στην αρχή, η προσέγγιση αυτή του να υπάρχει ένας και μόνο έλεγχος, αυτό είναι το καθαριστικό. Να είναι ανοιχτή η έλεγχη σε όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους, να υπάρχουν ε, απλές νομοθετικές διατάξεις για τις εκαθαρίσεις, να ε, γίνονται τυχαίοι ε, έλεγχοι από τυχαίους ελεγκτές, το να υπάρχει μία και μόνο ε, ένας και μόνος έλεγχο δεν σημαίνει ότι όλοι εμπιστεύονται όλους. Οι διεθνείς προδιαγραφές απαιτούν από όλους τους ελεγκτές να κάνουν την εργασία τους στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό ε, προϋποθέτει και την αξιολόγηση της ελεγκτικής εργασίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αξιολόγηση θα μας βοηθήσουν. Τα καλύτερα δεδομένα ε, προσφέρουν και καλύτερη κατανόηση, καλύτερη εποπτεία, προσφέρει τη δυνατότητα να εστιάζουμε την προσοχή μας στα αποτελέσματα. Και όταν μιλάμε για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι από αυτού, όπως είπε ήδη το 2014 η κυρία Λαπάγεβα σχετικά με την απαλλαγή του 2014. Όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι οφείλουν να έχουν συμφωνήσει το τι είναι η μία και νέα προσέγγιση. Ευχαριστούμε πολύ. Η εισαγωγή στο τρίτο τμήμα της συνεδρίασης αυτή ήταν ευχαριστώ πολύ. Οπότε ο επόμενος είναι η εισηγήτρια για την απαλλαγή του τελευταίου χρόνου η κυρία Παναγιώβα, η οποία είχε τις εμπειρίες της στον τομέα της επιμερισμένης διαχείρισης, όπως και ο κάθε εισηγητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί, αγαπητά μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ από την αρχή. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση για μένα και πιστέψτε με, εάν δεν είχα μια απο ακρόαση σχετικά με την προώθηση απόσπαση των εργαζομένων ε, θα βρισκόμουν εδώ. Και βρίσκομαι τώρα εδώ για την ανταλλαγή απόψεων με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και πιστεύω πως χρειαζόμαστε μία συνεργασία τον τομέα αυτό. Η διαχείριση δημοσιονομικών πόρων ίσως να μην είναι το πιο ελκυστικό ζήτημα προς ε, συζήτηση, αλλά οι πολίτες των χωρών μας σίγουρα το θεωρούν ε, υπατοστόχο σε εποχές υψηλής ενεργείας και έλλειψης πόρων και των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε η ατζέντα μας δεν περιορίζεται στην, στον καθορισμό του προπολογισμού της Ένωσης, αλλά όλα σχετίζονται με την πολιτική. Και αυτό το τονίζω επειδή όπως και το αντικείμενο της πρώτης συνεδρίας το απόγευμα, η γεωργία, η ανάπτυξη, όλα αυτά σχετίζονται με την πολιτική. Η διαχείριση των δημοσιονομικών είναι πολιτική και δεν πρέπει να ξεχνούμε τους στόχους των πολιτικών αυτών, τη βελτίωση της ζωής, της διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών. Λυπούμε που Περισσότερες από τις μισές εθνικές αρχές παρέλειψαν να συμμετάσχουν στην συνάντηση αυτή επειδή σύμφωνα με το άρθρο 317 της συνθήκης ο προϋπολογισμός της Ένωσης καταρτίζεται σε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και πιστεύω πως αποτελεί καθήκον μας να συνεργαζόμαστε μαζί και να διαχειριζόμαστε από κοινού τα δημοσιονομικά. Αυτό σημαίνει κατά την άποψή μου πως πρέπει να προσερχόμαστε στις αντίστοιχες συνεδριάσεις. Πρέπει να ελέγξουμε την δημοσιονομική επίδοση. Πρέπει να τονίσω κάτι το οποίο αναγκάστηκε να επαναλάβει το ελεγκτικό συνέδριο πως σε πολλές περιπτώσεις σφαλμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Εθνικές Αρχές, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν επαρκείς πληροφορίες ώστε να προλάβουν, να αποτρέψουν ή να διορθώσουν σφάλματα προτού προβούν σε δαπάνη χρημάτων. Γι' αυτό και θα επικεντρώσω στα εξής. Γιατί λοιπόν η Επιτροπή αυτή προσκάλεσε τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η Επιτροπή μας έχει το κύριο στόχο να ελέγξει πόσα χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, δηλαδή πόσα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται με βάση την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού συνοδρίου. Ήταν πάνω από 140 δισεκατομμύρια το 2015 είναι ένας, μέσο, ένας προϋπολογισμός μέσω μεγάλου μεγέθους, αν το συγκρίνει κανείς με τον προϋπολογισμό κάποιων κρατών μελών αλλά είναι μεγάλη σημασία για πολλά μικρά κράτη-μέλη, τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή είναι αυτή που σε τελική ανάλυση είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του προπολογισμού. Αλλά 80% των ενισχύσεων καταβάλλονται σε επιμερισμένη διαχείριση κυρίως στον τομέα της γεωργίας, της ε, περιφερειακής ανάπτυξης και της καταπολέμησης της ανεργίας. Κάθε χρόνο το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ε, παρατυπίες και σφάλματα κυρίως στην αγροτική, στις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης και συνοχής, που αποτελούν συχνά αποτέλεσμα ακατάλληλων ερμηνεών των κειμένων αυτό που βλέπουμε στο ελεγκτικό σύστημα των κρατών μελών, το λεγόμενο σύστημα πρώτου επίπεδου. Οπότε έχουμε μια έκθεση και σε αυτό το επίπεδο. Φυσικά και αν υπάρχουν προβλήματα από πλευρά των κρατών μελών, είναι φυσικό πως πρέπει να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη. Και οι φυσικοί συνομιλητές μας είναι τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο να ανταλλάξουμε απόψεις με όλους σας. Πέρυσι, όταν ήμουν εισηγήτρια για την απαλλαγή του 2014, δεν επιτύχαμε να έχουμε την ακρόαση αυτή. Προσκαλέσαμε κυβερνητικές αρχές, αλλά αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην συνάντηση. Φέτος, η Σλοβακική Προεδρία απέρριψε ευγενικά την πρόσκλησή μας και πιστεύω πως είναι ατυχές πως οι κυβερνητικές αρχές δεν προσέρχονται εφόσον ανησυχούν για τα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης. Πιστεύω πως αποτελεί ευθύνη των κρατών μέλων. Φυσικά και κάποια κράτη μέλη αποφασίζουν τα ίδια να τονίσουν, να ορίσουν ποιες είναι οι ευθύνες τους κατά την εφαρμογή του προπολογισμού μέσω κάποιων ειδικών δηλώσεων ορίζουν τις συναλλαγές υπό την εξουσία τους ως νόμιμες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φτάνει στο συμπέρασμα πως τα κράτη της Δανίας, της Σουηδίας και των κάτω χώρων αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη για τη χρήση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω δημοσίων εγγράφων. Αφετέρου, ο κοινων οι οικονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν πως τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να καταρτήσουν μια ετησία έκθεση. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας για τα ζητήματα αυτά, παρατηρήσεις και ίσως προτάσεις σχετικά με το ζήτημα των εθνικών διακηρύξεων ή δηλώσεων και τον ρόλο των κοινοβουλίων ως προς αυτό. Αλλά επίσης θα ήθελα να γνωρίσω τις απόψεις σας για τους μηχανισμούς ελέγχου πώς είναι οργανωμένοι στις χώρες σας, την ένταξή του, ενσωμάτωσή του στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει κάτι ως προς αυτό. Θα είχε ενδιαφέρον να συζητηθεί. Το άλλο ζήτημα είναι πως πρέπει φυσικά να διερωτηθούμε για τη φύση του διαλόγου που θέλουμε να προωθήσουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως ο διάλογος αυτός αποτελεί ζήτημα συνεργασίας και καλής βούλησης. Δεν υπάρχει ιεραρχία σε αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να βασίζεται σε μια ανταλλαγή ορθών πληροφοριών και σε απόλυτη αμοιβαία κατανόηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν βρίσκεται εδώ για να διδάξει, για να δώσει μαθήματα. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τα προβλήματα. Όταν το Ελεκτικό συμβούλιο, συνέδριο εντοπίζει σφάλματα στον τομέα της πολιτικής φυσικά και υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι και δικαιολογίες γι' αυτό. Αλλά εδώ βρισκόμαστε για να ακούσουμε ο ένας τον άλλον και για να καταδείξουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθνικές αρχές κατά την εφαρμογή του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μας γνωρίζουμε πως ε, μία από τις κύριες αιτίες για ε, για παρατυπίες είναι η περιπλοκότητα των κανόνων. Γνωρίζουμε πως από καιρό σε καιρό τα κράτη-μέλη όταν τα κράτη-μέλη καταρτίζουν τα ίδια κανόνες εφαρμογής, εκτελεστικούς κανόνες, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει το ίδιο. Για τον λόγο αυτό, είναι καλό κατά την άποψή μου τα ευτικά κοινοβούλια να εμπλέκονται όλο και περισσότερο στις διαδικασίες λήψης απόφασης έχουμε αυτή την ενδιαφέρουσα άσκηση που την ονομάζουμε απαλλαγή κάθε χρόνο. Αναρωτιέμαι πόσα μέλη, όχι εσείς που είστε οι, οι περί προϋπολογισμών, πόσα, θα αναρωτιέμαι πόσα μέλη του Κοινοβουλίου αυτού γνωρίζουν τι σημαίνει η απαλλαγή αυτή. Ακόμη και στις εθνικές και περιφερειακές αρχές για την εφαρμογή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη συνθήκη δεν ευθύνονται ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων αλλά λογοδοτούν μόνο στα δικά τους εθνικά κοινοβούλια. Και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποσκοπεί στο να δώσει μαθήματα. Η πολιτική δράση μας περιορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης και πρέπει να συνεργαστούμε με τα εθνικά κοινοβούλια. Γι' αυτό και ελπίζω τα εθνικά κοινοβούλια να υποστηρίξουν τη δράση μας, επειδή αποτελεί κοινό μας στόχο να, να παράσχουμε, να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη αξία για χρήματα και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Συμπεραίνοντα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να προτείνω τέσσερις δράσεις, τέσσερις προτάσεις συνεργασίας με σκοπό τη δημιουργία κάποιου βαθμού συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ζητήματα ελέγχου. Πάρτε τις προτάσεις αυτές ως μια πρώτη ιδέα ως, όπως θα τις έλεγα, δυνατές σκέψεις. Θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σας σχετικά με αυτές και πιστεύω πως ήταν χρήσιμο να αρχίζαμε από κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Η πρώτη μου πρόταση είναι πως η ετήσια παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου να γίνεται παρουσία των κοινοβουλίων. Φυσικά και θα ήταν ωραίο να γινόταν εδώ στι Βρυξέλλε. Είναι προφανέ πω η εφαρμογή του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Γι' αυτό και θα πρέπει να στοχαστούμε για τρόπους συνεργασία στο σημαντικό αυτό ζήτημα και να αρχίσουμε ήδη με την παρουσίαση τη ετήθεια έκθεση από κοινού. Από κοινού στην εταιρική αυτή σχέση. Η δεύτερη πρότασή μου είναι να προσπαθήσουμε στις συναντήσεις των επικεφαλής των επιτροπών ε, δημοσιονομικών του, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διοργανώνεται ένα εξάμεινο υπό την Προεδρία, συνήθως στη χώρα της Προεδρίας. Πιστεύω πως ένα συστηματικός τρόπος συνάντησης θα ήταν χρήσιμος για, και για τις δύο πλευρές. Η τρίτη πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου προσωπικού. Επειδή ως πολιτικοί γνωρίζουμε όλοι τι θα κάναμε χωρίς το προσωπικό μας. Και φυσικά αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο γραμματιών των εκαθοτε επιτροπών για να συζητούμε σχετικά με ψηφίσματα, συγκεκριμένα ζητήματα με τα κράτη-μέλη, αλλά επίση για τη διάδοση καλών πρακτικών. Παραδείγματο χάρη για την αποτροπή. Uh, in each parliament there could be a contact person in charge of transmitting this information. Και φυσικά η τελευταία πρόταση είναι εύκολη. είναι η συστηματική ενημέρωση των Εθνικών Κοινοβουλίων όταν η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στέλνει μια αποστολή στα κράτη-μέλη, που γίνεται από καιρό σε καιρό. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα να συζητήσω τις προτάσεις αυτές μαζί σας και ίσως μπορούμε να θεωρήσουμε την ακρόαση αυτή ως πρώτο βήμα για μια μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ε, και ίσως θα τον κόπο να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Αλανίσελε από τη Φονλανδία. Παλαιότερα ήταν ε, το φιλανδικό μέλος το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τώρα είναι αντιπρόεδρος ε, της αρμόδιας επιτροπής του στο κοινοβουλίο του. Κύριε Νίσελε, σας καλωσορίζουμε τορμά και έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση της σημερινής ε, συνάντησης για ένα σεμινάριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο μοντέλο για την χρηματοδότηση είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη ε, το σλόγγαν της ε, Χίλαρη Κλίντον, Stronger Together, πιο δυνατοί μαζί. Μπορούμε να είμαστε πιο δυνατοί μαζί. Έχω έξι σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Προηγουμένω ακούσαμε τέσσερα σημεία, τα δικά μου είναι έξι. Να σας πω καταρχήν πως είναι σημαντικό τα κοινοβούλια να έχουν λόγο στην λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Φιλανδία το δικό μας ε, κοινοβούλιο έχει μια ειδική επιτροπή η οποία πάντοτε ε, γνωμοδοτεί για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει να σας πω πως ε, πολλές φορές ακούμε και σχόλια επικριτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει και μια επιτροπή ελέγχου ενδεχομένω που θα αποτελεί ένα ανώτατο κοινοβουλευτικό όργανο, γιατί στην Φιλανδία ε, οι ελεγκτικές αυτές επιτροπές ε, έχουν την εποπτεία ε, επί των εθνικών λογαριασμών και αυτό κατοχυρώνεται μέσα από το είδο μας σύνταγμα. Πρέπει να σας πω πως λαμβάνουμε κάθε χρόνο την έκθεση της του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και νομίζω ότι η δήλωση που γίνεται για τα θέματα αυτά θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν και τους ε, μηχανισμούς ε, σταθερότητας όπως επίσης και όλα τα σχετικά με το ESM ζητήματα. Να σας πω επίσης πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναγνωρίζουμε και να γνωρίζουμε τα συμπεράσματα της έκθεσης της, ε, του Ελληνικού συνεδρίου και πρέπει να σας πω πως η έκθεση αυτή δεν είναι η μόνη, θα πρέπει και οι ειδικέ εκθέσεις του Ελληνικού συνεδρίου να λαμβάνονται υπόψη, γιατί τα συμπεράσματα και τα ευρήματα μας βοηθούν στο να αξιολογήσουμε την ποιότητα που έχει η διαχείριση που γίνεται των ευρωπαϊκών κονδυλίων και ο τρόπος με τον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί και πού ακριβώς βρίσκονται οι κίνδυνοι για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τι λέει η εκθέση του ελεγκτικού συνεδρίου, πως εάν τα κράτη-μέλη, οι αρχές τους, οι ανεξάρτητοι ελεγκτές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, θα μπορούσαν να έχουν προλάβει ή ανοιχνεύσει ή διορθώσει ένα σημαντικό αριθμό των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν. Άρα λοιπόν και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε κατά νου. Τέταρτο. Καταλογισμοί. Ένα θέμα στο οποίο δεν αναφέρεται η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, δηλαδή πώς μπορεί η διορθωτική δράση να λαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, αυτή η ευθύνη του να ληφθεί δράση θα πρέπει να βαρύνει τον Υπουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνο για αυτήν την πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Άρα λοιπόν η ανάγκη υπάρχει και θα πρέπει αυτά τα συμπεράσματα και οι εκθέσεις του ε- Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου να λαμβάνονται πιο πολύ υπόψη και σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι τα όσα γίνονται σήμερα δεν είναι αρκετά θα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις των καταλογισμών που επιβάλλονται και σε κάποιους κλάδους της οικονομίας, γιατί ξέρετε πως υπάρχει ο ηθικός κίνδυνος αυτή τη στιγμή. να πληγούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αυτό έγινε με τον κατάλληλο τρόπο. Το πέμπτο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι ίσως χρειάζονται περισσότεροι ε, έλεγχοι που θα γίνονται παραλίλω, δηλαδή μεταξύ εθνικών ελεγκτικών αρχών από τα ε, κοινοτικά όργανα για να βλέπουμε ακριβώς την πορεία ε, που ακολουθούν αυτά τα διαφθορτικά ταμεία. Να παρακολουθούμε λοιπόν τη δαπάνη, τον τρόπο με τον οποίο ε, γίνεται σε όλη την Ευρώπη, πώς τη διαχειρίζονται οι αρχές και αυτές οι παράλληλες εκθέσεις θα μας προσφέρει αρκετή γνώση που θα μας επιτρέψει να επιλέξουμε αργότερα τα κατάλληλα εργαλεία για τις διορθωτικές πολιτικές. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε στον κλάδο αυτό να συνεργαστούμε μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και βεβαίως πάντα με την ε, συμβολή των Εθνικών Αρχών. Επίσης, τελευταία μου παρατήρηση, τι χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε ε, πιο εφάνταστοι και πρέπει αυτά που κάνουμε να εφαρμόζονται καλύτερα στην πράξη, να έχουμε βελτιωμένα, ε, βελτιωμένες επιδόσεις στην εφαρμογή. Λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερο διοικητικό βάρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε ανάλυση κινδύνου και οι έλεγχοι να γίνονται σύμφωνα με αυτή την ανάλυση. Όταν λοιπόν οι διοικητικέ διαδικασίε γίνονται με σωστό τρόπο στα κράτη-μέλη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε του ελέγχου με τον τρόπο αυτό που σας προτείνω. Και αν γίνονται λιγότεροι έλεγχοι θα είναι λιγότερο και το διοικητικό βάρος. Να σας πω πως ε, στην Φιλανδία προσπαθούμε να μειώσουμε ε, την ε, αχρίαστη γραφειοκρατία και νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά. Θα κλείσω λοιπόν με το εξή συμπέρασμα. Οι νέες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέματα της διαχείρισης με τους νέες ευθύνες που θα βαρύνουν και τις εθνικές ελεγκτικές αρχές αλλά και τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει για να κάνουν τη διαφορά να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτό με έναν αποτελεσματικό τρόπο και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι με τα όσα παρουσιάστηκαν στο σημείωμα το ενημερωτικό για αυτή την συνάντηση όπου είπε όλοι πως η κοινοβουλευτική εποπτεία θα πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα εργαλεία και με όλους τους τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε να επηρεάσουμε και την απόδοση και την εφαρμογή όλων των συστημάτων και των οργάνων που ε, μπλέκονται στην ε, διαχείριση ε, και στην δαπάνη των κοινωτικών κονδυλίων. Ακόμα περισσότερο θέλω να σταθώ e Θέλω να σταθώ λοιπόν στο γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και για να τα λύσουμε σε εθνικό επίπεδο πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες, χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, χρειαζόμαστε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Νομίζω πως θα πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν περαιτέρω. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι τα εθνικά κοινοβούλια να γνωρίζουν ποια είναι τα βασικά ευρήματα των εκθέσεων του ελεγκτικού συνεδρίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, έτσι ώστε να γνωρίζουν ποιες είναι οι διορθωτικές κινήσεις που γίνονται σε εθνικό επίπεδο και πώς επηρεάζουν τους δικαιούχους. Um, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και να σας πω πως ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια αντίστοιχη συζήτηση και κάποια άλλη στιγμή τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ε, Βεβαίω, ε, διερωτώμεθα τι είναι το καλύτερο. Ε, πώς να παραμείνουμε μεταξύ μας σε επαφή. Ε, έχουμε συζητήσει με τα Εθνικά Κοινοβούλια και πολλές φορές ε, όλοι μας τιμώναμε γιατί δεν γινόταν τίποτα. Εντάξει, ερχόμαστε εδώ, τα λέγαμε και μετά πηγαίνουν όλοι σπίτι τους και τίποτα. Τώρα όμως θέλουμε πραγματικά να έχουμε έναν ουσιαστικό διάλογο. Γιατί ε, το ευρωπαϊκό επίπεδο το εχθρεύονται πάρα πολύ πολλά κράτη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει έτσι κάποια εχθρότητα εναντί των κρατών μελών. Μόνο που εσείς έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε και μπορείτε να τα καταφέρετε πολύ καλύτερα παρεμβαίνοντας την κοινή γνώμη από ότι εμείς. Κάπως πρέπει να λυθεί όλο αυτό το θέμα και πρέπει να γίνει κατανοητό το γιατί γίνονται όλα αυτά. Ε, ξέρετε και σήμερα μιλάμε, όχι απλά για να μιλάμε μέχρι να γίνει η δεξίωση, αλλά γιατί πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Να βοηθήσουμε εσάς, ε, τα κράτη-μέλη, να επιτύχετε πολλά πράγματα. Έγινε νομίζω κατανοητό από όλου ότι πρέπει να ενισχυθεί η ε, συζήτηση, ο διάλογος. Ε, χαίρομαι που ο κύριος Κίρστενς από τη Λετωνία επιθυμεί να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου σε αυτά που είπε ο Φινλανδός συνάδελφος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του ως προς το ότι τα Εθνικά Κοινοβουλία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Αυτό που δεν συζητήθηκε είναι η αλλαγή της ε, πολιτικής ε, κατάστασης σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία. Ας πάμε στη Λετωνία. Έχουμε έναν οργανισμό πληρωμών που ελέγχει την χρήση των κονδυλίων. Υπάρχουμε και έχουμε και έναν έχουμε μια σχετική επιτροπή στο Κοινοβούλιο που και αυτοί κάνουν το ίδιο και το ελεγκτικό συνέδριο. Όλοι αυτοί ελέγχουν τις ε, γεωργικές ε, δαπάνες Δυστυχώς όμως πάρα πολλά έχουν υποβαθμιστεί λόγω των εξελίξεων στη, στη Ρωσία. Ξέρετε, εμείς είμαστε τα μεγαλύτερα θύματα. Έχουμε τρία λιμάνια. Και τι έγινε. Ε, οι διασυνδέσεις ε, ήταν προσανατολισμένες ανατολικά και δυτικά και μετά τις εξελίξεις ε, στην Ουκρανία η ανταλλαγή εμπορευμάτων με τη χώρα αυτή μειώθηκε και το ίδιο συνέβη βέβαια και με τον όγκο συναλλαγών στα λιμάνια μας. Ε, τος χάρη, στο λιμάνι της Ρήγας είχαν λάβει χώρα ε, βελτιτικές εγκαταστάσεις για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση. Ε, επειδή λοιπόν η ε, ήταν πάρα πολύ μεγάλος όγκος συναλλαγών με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μετά τις αλλαγές προέκυψε ένα πρόβλημα. Εμείς είχαμε αναγκαστεί να αγοράσουμε μηχανήματα, ε, μηχανές σκάνερ. Τα είχαμε αγοράσει όλα αυτά, την απαραίτητη υποδομή. Τώρα πια όμως δεν είμαστε κέντρο διαμετακόμισης εμπορευμάτων. Και τι συμβαίνει, μας λένε οι Ευρωπαίοι ότι δεπανήθηκαν όλα αυτά τα κονδύλια, από την άλλη όμως δεν ελείπτει υπόψη, δεν ελείψαν υπόψη οι πολιτικές εξελίξεις. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Χρησιμοποίησαμε τα παρέτα κονδύλια, τώρα όμως οι υποδομές δεν την χάνουν χρήσης και συμφωνώ μαζί σας ότι και η διοίκηση αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Εμείς είμαστε ένα μικρό κράτος, βρισκόμαστε δίπλα σε έναν οικονομικό γίγαντα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να το λάβει αυτό υπόψη της. Εμείς ε, επηρεαζόμαστε περισσότερο από τις πολιτικές εξελίξεις. Και νομίζω ότι οι Βρυξέλλες δεν το κατανοούν αυτό σωστά. Ε, επιβλήθηκαν κυρώσεις. Αυτές οι κυρώσεις ίσως να μην αφορούν τόσο τη Γερμανία, αλλά στις χώρες της Βαλτικής ε, οι εξαγωγές γάλακτος καταστράφηκαν, κατέρευσαν. Σας είπα, ε, δημιουργήσαμε υποδομή με ευρωπαϊκά κονδύλια, τώρα όμως αυτή η υποδομή λόγω των ε, πολιτικών εξελίξεων είναι άχρηστη, δεν χρησιμοποιείται. Εξάλλου πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και για, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε εμεί πάρα πολύ που φέρατε στη συζήτηση ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχαμε κατά νου και πολύ δίκαια περιγράφεται έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και στη συνέχεια τοποθετούνται κάποια εργοστάσια εκεί και οι εξαγωγές καταραίουν. Είναι προβλήματα με τα οποία αγωνιζόμαστε όλοι μας αλλά πιστεύω πως πρέπει πάντα να προσμένουμε τα, τα πάντα, αλλά πρέπει παράλληλα επίσης να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά. Σήμερα τα προβλήματα είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν από πέντε χρόνια, για να μην μιλήσουμε με το πώς ήταν πριν από 13 χρόνια όταν ήρθα εγώ. Τότε ασχολούμασταν με εντελώς διαφορετικά πράγματα. Από την οπτική γωνία του σήμερα, το παρελθόν μπορεί να μοιάζει σαν τους παλιούς καλούς καιρούς και τους καιρούς εκείνους, όπου το, όπου το αντικείμενο των συζητήσεων ήταν σχετικά μικρά προβλήματα. Γι' αυτό και η ανταλλαγή απόψεων είναι πολύ σημαντική και, το ζήτημα το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο, πώς θα βελτιώσουμε τον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Αν κοιτάξουμε τα προγράμματα αυτά σήμερα, είναι να σου σηκώνεται η τρίχα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ξανακαταστήσουμε φυσιολογικό τον κόσμο και αυτό πιστεύω δεν θα κοστίσει πάρα πολλά χρήματα. Θέλω να ρωτήσω τον Αλάν Ίσελιν πως βλέπετε την κατάσταση επειδή στο δημοσιονομικό έλεγχο εμείς πάντα διαπιστώνουμε πως καταραίει ο κόσμος μας ή μάλλον ότι διαιρείται μεταξύ χωρών δοτών και χωρών παραλειπτών. Οι παραλήπτες πάντα θεωρούν ότι λαμβάνουν πολύ λίγα, οι δότες ότι δίνουν πάρα πολλά Οπότε από την άποψή σας, πώς θα τα καταφέρουμε να παρακινήσουμε όλες, όλα τα κράτη-μέλη σε μια δίκαιη κατανομή πόρων, επειδή πιστεύουμε πως, αυτό, πως υπάρχουν εκεί διαφορές συμφερόντων, αλλά και διαφορές πρόσληψης, αντίληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εκάστοτε κράτη-μέλη. Πιστεύω πως ε, σε κάθε κράτος μέλος η η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ίδια, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ως αντικείμενο τα χρήματα, αλλά τα κοινά στοιχεία. Οπότε θα σας παρακαλούσα να προβείτε σε μια σύντομη τοποθέτηση. Καλή ερώτηση θα έλεγα. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το ότι στα κράτη-μέλη τα εθνικά κοινοβούλια έχουν έναν αδύναμο ρόλο στα, για τα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια. Αυτός πρέπει να ενδυναμωθεί σε επίπεδο κρατών μέλων. Η καλύτερη συνεργασία σε δια της οδού της επιμερισμένης διαχείρισης πιστεύω πως απασχολεί επίσης το Συμβούλιο. Το αντιλαμβάνομαι σχετικά συχνά κατά τη σύνοδο του ΕΚΟΦΗΝ. Εκεί όλο αυτό δεν είναι κάποιο μεγάλο ζήτημα ενώ θα έπρεπε να, να δοθεί περισσότερη προσοχή. Θα μπορούσαμε να πούμε στους υπουργούς μας, κοιτάξτε, πρέπει να εξετάσουμε το ζήτημα αυτό όταν διαπραγματευόμαστε με το ελεκτικό συνέδριο στις συναντήσεις. τα κράτη-μέλη μπορούν επίσης να κάνουν το δικό τους μερίδιο στην εργασία. Πιστεύω πως είναι σημαντικό πως η εργασία πρέπει να γίνει σωστά σε επίπεδο κράτους μέλους και σε επίπεδο αποφελούμενων. Επειδή σε διαφορετική περίπτωση δεν θα επιτύχουμε επαρκείς βελτιώσεις. Ο κύριο ε, Λαζάρου μου είπε ότι πήγε στο Συμβούλιο και πρέπει να περιμένει τέσσερι ώρε για το ΕΚΟΦΗΝ. Και διερωτώ με το Συμβούλιο ενδιαφέρεται για τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μπορείτε να μα απαντήσετε σε αυτό. θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να ενδιαφέρονται για το τι κάνει το Ελληνικό συνέδριο. Τουλάχιστον στο επίπεδο της απόδοσης, νομίζω πως θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται να αποφασίσουν εκ των προτέρων ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιες είναι οι επιπτώσεις που επιδιώκουν μέσω των προτάσεων κάποιου έργου στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να έχει κάποιες κοινέ καθεντήριες γραμμές για όλα τα κράτη-μέλη για να μπορούν να εγκρίνουν ε, ή να υιοθετήσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές επιταγές και στόχους που έχουμε στις ε, στρατηγικές για τα δίκτυα, για παράδειγμα. Γιατί πρέπει να σας πω πως η έκθεση δική μας λέει πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευθυγράμμιση μεταξύ της στρατηγικής του 2020, και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών μελών. Παρόλα τα σύμφωνα εταιρικής σχέσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσουν εκ των προτέρων ποιες ή μάλλον ποιοι είναι οι στοχευμένες, ποιες είναι οι στοχευμένες προτεραιότητες τουλάχιστον στα έργα τα οποία θα τύχουν συγχρηματοδότησης. Ήγκη και η ώρα της αλήθειας, λέει η πρόεδρος. Και ε, φτάνουμε την ε, τελευταία εισηγητή. Ματίνα, τι μένει από τη <laughs> διαχείριση και τι πρέπει να ε, λάβουν υπόψη συνάδελφοι ε, πριν φύγουν και πριν δώσουμε το λόγο στον τελικό ζητητή, τον κύριο Τσέλερ. Κοιτάξτε, το πιο σημαντικό που θα πρέπει να παραμείνει ως ε, μήνυμα είναι ε, δεν είναι η τελευταία φορά που έχετε κανείς εδώ σε ακρόση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι συγητές πρέπει να μιλάνε ανοιχτά για τα προβλήματα, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που τουλάχιστον πέρσι δεν το άκουσα, ε, μου έλειψε. Και ως εκ τούτου ζηλεύω τον συνάδελφό μου τον κύριο Τσέλα, ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα πριν συντάξει την έκθεσή του να μιλήσει με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ως εκ τούτου να μην αλλάξει κατάσταση, να ξανάρθουμε του χρόνου Βλέπετε ότι εμείς είμαστε συμπατικοί άνθρωποι και είμαστε ανοιχτοί και για συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ούτε και εμείς δαγκώνουμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο στον ε, κύριο Τσέλα, τον εισηγητή για την κατακλίδα των εργασιών μας ε, και μετά ε, έχουμε προβλέψει δεξίωση στο δεύτερο όροφο. Είσαστε όλοι καλεσμένοι. Ξέρετε ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθετε Ε, επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα του Ευρωπαίου Οικονομικού Εισαγγελέα και υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις ε, των κρατών μελών. Εμείς ε, προσπαθήσαμε να ε, έχουμε κάτι το οποίο όμως θα προστατεύει καλύτερα τον ευρωπαϊκό προευλογισμό από τις απάτες. Μέχρι τώρα μερικές φορές δεν ήμασταν σίγουροι ότι οι οικονομικές ε, υπηρεσίε αρμόδιες εισαγγελείς ε, των κρατομελών θα δραστηριοποιούνταν οποτεδήποτε προέκυπταν απάτες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαίο οικονομικό εισαγγελέα. Τον χρειαζόμαστε αυτόν. Ε, ο οποίο ασχολείται και με τους προπολογισμού των κρατών μελών. Βεβαίω τώρα φοβόμαστε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα διαφωνήσουν, δικαιωμά βέβαια είναι αυτό, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλές φορές έχουμε δυσκολίες να ε, εγκριθούν προϋπολογισμοί υπολογισμοί κρατών μελών που είναι ακριβώ εκείνα τα κράτη-μέλη που διαφωνούν για τον οικονομικό εισαγγελέα. Ε, Υπάρχει κάποια σχέση, αν θέλετε, ανάμεσα στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων αφενός και την ε, παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, αφετέρου. Ε, μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα για το ότι δεν μπορεί κανείς να δείξει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, στις οικονομικές αρχές των κρατών μελών. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τσέλλερ, ο οποίος ε, όπως σα είπα θα κλείσει τη συνεδρία. ευχαριστώ όμως όλους σας που ήρθατε. Ευχαριστώ τη Γραμματεία για την οργάνωση της ε, σημερινής δύσκολης συνάντηση. Κύριε Τσέλλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην ε, Γερμανία πολύ συχνά λέμε και εμείς κάθε αρχή και δύσκολη. Και έτσι λοιπόν πράγματι εσείς που είστε οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Περιφερειών, ήρθατε σήμερα εδώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου Προπληγισμών. Δεν ήταν εύκολο αυτό, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία. Εγώ λυπάμαι πολύ που ε, συνάδελφοι της Επιτροπής Ελέγχου Προπληγισμών ήταν παρόντες. Δεν ήταν βέβαια και όλοι όσοι θα επιθυμούσα, αλλά εκείνο που μου έλειψε ήταν το ότι δεν ήταν εδώ οι συνάδελφοι εκείνοι που είναι σημαντικοί για τα θέματα που συζητάμε. Δηλαδή ο αρμόδιος για θέματα περιφερειών, για θέματα γεωργίας. Αυτοί όλοι ζητάνε συνεχώς αδιάλειπτα να συνεργαζόμαστε με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά τελικά δεν ήρθαν σήμερα εδώ. Πάντως, εντάξει, μπας περιπτώσει, θα βελτιωθεί η κατάσταση, ε, θα τους ασκήσουμε πίεση, ε, γιατί όλοι επιθυμούμε να υπάρχει αποτελεσματική χρήση κονδυλίων στο πλαίσιο του χρονικού πλαισίου που μόνοι μας έχουμε θέσει. Κατά τα άλλα, νομίζω κατέστη απόλυτα σαφές ότι τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα στις περιφέρειες και κυρίως στις περιφέρειες εκείνες ε, οι οποίες φέρουν ευθύνε. Αντιμετωπίζονται αυτά ως ε, ένα εργαλείο το οποίο κατά τα άλλα δεν θα τους προσεφέρετο. Ε, βεβαίως ε, τα κονδύλια δεν είναι αυτονόητα, δεν είναι δεδομένα, δεν είναι χριστουγεννιάτικο δώρο που το βρίσκει κανεί κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όχι, πρέπει κανεί να προετοιμαστεί, ε, να δείξει ενδιαφέρον για τα κονδύλια αυτά για να μπορούν να τα λάβουν οι περιφέρειες και επίσης ε, και για να μπορούν να συμμετέχουν και στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Επειδή λοιπόν ελέγχεται επανειλημμένα ότι και τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά κονδύλια είναι περιορισμένα, ακροθυγώς ε, τέθηκε το θέμα του Brexit. Αν τελικά υπάρξει Brexit, δηλαδή αποχωρήσει μία από τις ε, μεγάλες χώρες ε, συνεισφορής στον ευρωπαϊκό προβλησμό, θα, ε, θα ξανατεθεί το θέμα αναδιάταξης του προϋπολογισμού, του ευρωπαϊκού, του ανοσιακού προϋπολογισμού. Θα δούμε και εμείς τα εργαλεία που θα έχουμε τότε στη διάθεσή μας, γιατί το σημαντικότερο είναι να δούμε κατά πόσον ε, μπορούμε να προχωρήσουμε με τον ευρωπαϊκό, τον ενωσιακό προβλησμό. Επ' αυτού χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Νομίζω ότι η αρχή έγινε. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαν ε, αρκετοί συνάδελφοι στις Βρυξέλλες και ελπίζω ο διάλογος που ξεκίνησε σήμερα να συνεχιστεί και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Η συνεδρίαση έκλεισε. Ελάτε στη δεξίωση στο δεύτερο όροφο. Ευχαριστώ πολύ.